Good afternoon everybody. I think... Καλησπέρα σας λέει ο πρόεδρος. Ας αρχίσουμε την συνεδρίασή μας. Για πρώτη φορά προεδρεύω στην Επιτροπή Απασχολήσεως, αλλά θα το πράξω με μεγάλη χαρά και είναι τιμή μου να προεδρεύσω σε αυτήν την ε, σημαντική συνάντηση, να βλέπω όλους ε, εσάς ε, τους χαμογελαστούς όπως και τους συναδέλφους ε, διερμηνείς είναι κάτι το πολύ ευχάριστο. Για να δούμε όμως τα της ημερησίας διατάξεως. Πρώτα πρώτα, σας ερωτώ, υπάρχει ε, κάποια ένσταση για την ημερησία διάταξη. Εάν όχι, τότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Τέλεια. Επίσης, θα πρέπει κάτι να σας πω όσον αφορά τις αγγελίες του Προέδρου. Έχουμε διερμηνία από όλες τις γλώσσες. Και έχουμε πλούσιο γλωσσικό προφίλ, έχουμε και... Ε, δεν έχουμε, συγγνώμη, μόνο τα μαλτέζικα. Και επίσης θα πρέπει να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους. Τον Ανδρέα Μποξούρ, την Ανδρέα Μποξούρ από την Ουγγαρία, ε, Λέξμαν από την Ουγγαρία, επίσης την ε, Ελέν Φριτζόν από την Σουηδία, την Ντομινίκ Μπίλντ από την Γαλλία και τελευταία αλλά σημαντική την Μαργαρίτα Δελαπίσα Καριόν από την Ισπανία και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλή συνεργασία στο μέλλον. Και τώρα προχωρούμε στην μερσία διάταξη. Θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά προηγουμένων συνεδριάσεων και να έχουμε μία ώρα για τα σχετικά με την έκθεση του Eurofound για την παινία, για την φτώχεια, στην απασχόληση, στην, στους χώρους ε, της εργασίας. Ήδη ε, έχουμε συνοηθεί, έχουμε συντηθεί, ξέρω ότι είναι δουλειά σας, ε, κυρία Ντάφνη Άρεντ που είστε προϊσταμένοι μάνατζερ έρευνας του Eurofund και θα μας ε, παρουσιάσετε σε γενικές γραμμές πώς εξελίχθηκε αυτό το πρόβλημα αυτής της ε, φτώχειας κατόπιν της χρηματοοικονομικής κρίσεως το 2008 και τις επιπτώσεις όσον αφορά ε, την κατάσταση των Ευρωπαίων. Πρόκειται να βασιστείτε, για αυτή σας την παρουσίασετε, στην έκθεση του 10 ε, του Eurofound, επ' αυτού του θέματος, αλλά θα μας ενημερώσετε με πρόσφατα στοιχεία ε, τα οποία ετοιμάσατε ειδικά για τη σημερινή παρουσίαση. Έχετε για 10 λεπτά τον λόγο και στη συνέχεια ε, θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή για μένα και για την Eurofound να είμαι σήμερα εδώ και να μπορέσω να σας παρουσιάσω ε, την μελέτη μας αυτή για την φτώχεια των εργαζομένων. Έχουμε 20 εκατομμύρια, όπως ξέρετε, εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ε, εισόδημα για το νοικοκυριό τους κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Αυτό σας το λέω γιατί πρόκειται για τον αριθμό που είχε τεθεί από την Ευρώπη από εμά στα πλαίσια της του 2020. Θέλαμε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια να σωθούν από τον κίνδυνο της ε, ε, περιθωριοποίησης και της φτώχειας. Οπότε αξίζει το θέμα της προσοχής των κέντρων αποφάσεων το ότι έχουν απασχόληση επομένω δεν αρκεί, γιατί χρειάζονται ποιοτικέ θέσει εργασία, χρειάζεται κοινωνική πρόνοια, ακριβώ όπω προβλέπει ο κοινωνικό πυλώνα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, που είναι νομίζω ε, στέγανο και θα επανέλθουμε σε αυτό. Και ε, από το 2010 έχουμε ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε το 2017 ε, κάποια έκθεσή μας που δημιουργήθηκε και θέλουμε τώρα να δώσουμε συνέχεια στη μελέτη αυτή για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα κατά την κρίση. Και όπως μας ε, ζητήσατε έχουμε επικαιροποίησει αυτά τα στοιχεία από το 14, το 17 και το 18 και όπως βλέπετε σε αυτή την διαφάνεια ε, κάποια από αυτά τα στοιχεία και κάποια από τα συμπεράσματά μας για να δείτε ακριβώς ε, τι γίνεται ε, από πλευράς κοινωνικής για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτό το πρόβλημα. Στην παρουσίασή μου θα σας πω τι γίνεται για κάποιους εργαζομένους μερικής απασχόλησης κάποιους που ασχολούνται με ε, θελοντική εργασία, με αυτό αυτοαπασχολούμενους, ε, ε, που είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από αυτό το φαινόμενο. Βλέπετε τώρα στην επόμενη διαφάνεια ότι έχουμε ε, τρεις-τέσσερις βασικές αιτίες. Πρώτα-πρώτα έχουμε χαμηλή αμοιβή ε, και λέμε ότι δεν είναι αυτό η βασική αιτία του φαινομένου, αλλά επειδή ακριβώς έχουν ε, πολύ μικρή αμοιβή, αυξάνεται πάρα πολύ ο κίνδυνος να πέσουν σε αυτήν την ε, παινία. Γιατί πολλές φορές αυτός ο κίνδυνος εξαρτάται βέβαια και από τη σύνθεση του νοικοκυριού τους. Οπότε, αν κάποιος που έχει χαμηλό μισθό ή ημερομίσθιο έχει και πρόσωπα που από αυτόν, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό και οι μονογονικές οικογένειες ε, τόσο πολύ κινδυνεύουν ε, γιατί εξορισμού έχουν ε, εισόδημα μόνο από μία πηγή. Και επίση όταν υπάρχουν πολλοί κατιόντες και αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος και για οικογένειες με πατέρα και μητέρα και επίσης όταν υπάρχει σχέση απασχόληση ή απασχόληση χαμηλής εντάσεως στη, στο νοικοκυριό. Και επίσης όταν ακριβώς υπάρχουν πολλά παιδιά που εξαρτώνται από τους γονείς είναι υψηλές οι ανάγκες του νοικοκυριού και άρα υψηλός και ο κίνδυνος. Και όπως αναφέραμε ε, για την περίπτωση των μονεγών οικογενειών και μεγάλων οικογενειών ε, αυτοί κινδυνεύουν και αυτό ισχύει για τα νοικοκυριά όπου έχουμε ας πούμε δύο ενήλικες που πήγαν να μείνουν με τους γονείς τους και θα δούμε μετά για ποιες ομάδες προσώπων μιλούμε ε, και για κάποιους που χωρίς να θέλουν δουλεύουν σε ενεργή απασχόληση, αυτοπασχολούμενους χωρίς να έχουν υπαλλήλους και επίσης αυτοί που έχουν κάποια προσωρινή σύμβαση εργασία. Είναι κατηγορίε που αναφέρουν προηγούμενο Και για να δούμε επίση μια γενική έποψη του φαινομένου, όπω έχουν τα πράγματα και όπω έχουμε ενώσει τα στοιχεία μα ε, επί τη βάση του 18. Βλέπετε ε, ότι είναι ε, μικρέ οι μεταβολέ, 9,4% έχουμε σύμφωνα με τα στοιχεία του συνόλου της Ένωσης για το 17 Οπότε ένας στους δέκα περίπου από τους εργαζομένους ε, έχει κίνδυνο τέτοια ασπενίας. Όμως υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των χωρών. Πώς βλέπετε σε αυτό το γράφημα έχουμε αλλαγές ε, σε κάθε περίοδο 14, 7 μάλλον 14-18 τα στοιχεία που έχουν από αυτέ τι χώρε. Για κάποιε χώρε λοιπόν είναι τα στοιχεία και από το 17. Όταν βλέπετε αυτό το χοντρό βέλο σημαίνει ότι η αλλαγή κατά την περίοδο καταμέτρησης είναι μεγάλη και ε, είναι τα τελευταία χρόνια, ενώ αν δείτε αντίστοιχα ένα λεπτό βέλος, είναι η διαφορά ε, πιο παλιά, για όλη, της, για όλη την περίοδο 7 έως ε, τώρα. Λουξεμβούργο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται στην ελληνική, στη διατροφή, ε, σε ξενοδοχεία. Έχουν εκεί κάποια συγκεκριμένη ελάχιστη αμοιβή ή ημερομίσθιο και αυτό το αναφέρουμε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς εργαζομένους και γι' αυτό εδώ βλέπουμε υψηλό ποσοστό, πολύ υψηλό ποσοστό. Επίσης, αξίζει να παρατηρήσουμε τι γίνεται στην Ρουμανία που έχει το υψηλότερο ποσοστό ακόμη όσον αφορά αυτού του είδους την ε, παινία. Ε, αυτά το 16 όμως δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών στην Ήπεθρο, ε, δηλαδή για κάποιους που δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν δεξιότητες, ε, ε, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Μετά, Γαλλία, Γερμανία, κάτω χώρες, Αυστρία, χώρες της Επιρροτικής Ευρώπης, εδώ έχουμε στεγανές συλλογικέ συμβάσεις και εδώ βλέπουμε χαμηλά ποσοστά. Όμως αυτό δεν ισχύει για μη κλασικούς παραδοσιακούς, παραδοσιακές μορφές εργασίας. Υπάρχει δηλαδή πλαίσιο προστασία για τους πλήρως απασχολουμένους, αλλά όχι για τις μη παραδοσιακές μορφές εργασίας, απασχόλησης. Παρακάτω τώρα, για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα για διάφορες μορφές, διάφορα είδη σύμβαση εργασίας, όπως βλέπετε στο γράφημα, η πλήρους απασχόλησης και οι μόνιμες διαρκείς σύμβαση εργασίας είναι αυτοί που έχουν ε, τον μικρότερο κίνδυνο για τέτοιου είδους φτώχεια. Και βλέπουμε εδώ αυτές τις επτά στήλες και Βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ διαφόρων μορφών απασχόληση, ε, εθελούσια, ακούσια κλπ. Ε, όλα αυτά κατόπιν δηλώσει των δύο των ε, εργαζομένων. Δηλαδή ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ προσωρινής σύμβασης που, και, και, και αυτών που χωρίς να θέλουν δουλεύουν, δουλεύουν σε μερική απασχόληση γιατί δεν μπορούν να βρουν περισσότερες ώρες απασχόλησης και αυτοί επομένως ε, κινδυνεύουν πάρα πολύ και θα πρέπει να μην ξεχνούμε Βέβαια 48% είναι για τους ε, ανέργους, υψηλότερο ποστό, αλλά ήδη το 30% που βλέπουμε εδώ ήδη είναι υψηλό. Άρα προσωρινή απασχόληση μη τυπικός κλασικός τόπος εργασίας, συγκεκριμένη ε, περίοδος απασχόλησης, υπάρχει κίνδυνος. Πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μια διαρκή σύμβαση, μετά έχουν τους αυτοαπασχολούμενους. Εδώ είναι δύσκολη περίπτωση τούτο και θα επανέλθουμε γιατί σε κάποιες χώρες, σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους εποχιακούς εργαζομένους. Πού σε κάποιες περιπτώσεις ε, κατατάσσονται στους αυτοπασχολούμενους. Άλλο θα πει, προσωρινή απασχόληση ε, και μερική απασχόληση. Εκεί είναι ο κίνδυνος και γι' αυτό αυτοί είναι αντίστοιχα οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο. Για να δούμε τώρα ε, αυτούς που έχουν μερική απασχόληση. αποκλήσεις μεταξύ των χωρών 4% στη Δανία και 42% στην Βουλγαρία και σε κάποιες χώρες ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και από τους πλήρους απασχόλησης. Σε... Κάτω χώρες και Δανία είναι ίδιος ο κίνδυνος. Και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το πώς γίνεται η μέτρηση και τι ορισμός δίνεται για αυτού του είδους την φτώχεια. Γιατί όταν πριν είδαμε τα συνολικά στοιχεία είδαμε ότι το ποστό για την Ένωση είναι το συνολικό και επομένως κάποιος θα πρέπει να έχει δουλέψει τουλάχιστον 7 μήνες τη χρονιά για να υπολογιστεί. Αλλά όμως όσον αφορά το εισόδημα του νοικοκυριού μετράτε το μέσο εισόδημα που θα πρέπει να είναι κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος για να θεωρηθεί ότι το εν λόγω νοικοκυριό ή το εν λόγω πρόσωπο κινδυνεύει. Επίσης πάμε ταχαίως στα θέματα Α, είπαμε για, τα, για τις αιτίε, είπαμε ότι είναι η σύνθεση, η σύνθεση του νοικοκυριού για αυτή τη μορφή φτώχεια. Σε χώρε όπω τι κατοχώρε, διαπιστώνουμε ότι έχουν μερική απασχόληση είναι ε, το βασικό εισόδημα του νοικοκυριού, οπότε υπάρχει λιγότερος κίνδυνος τέτοιας φτώχειας. Επιστρέφουμε τώρα στους ε, μερικές απασχόλησης εργαζομένους συνολικά κινδυνεύουν περισσότερο σε χώρες όπου συνδυάζονται διαφορετικές μεταβλητές, δηλαδή μικρότερη αμοιβή, ε, μη σταθερή δουλειά, ε, εξαρτώμενα μέλη του νοικοκυριού, ε, συγκεκριμένη δομή της εργασίας τους. Τώρα, έχουμε αυτούς που χωρίς να θέλουν έχουν μερική απασχόληση. Κατά την κρίση, επειδή είχαμε πτώση της απασχόλησης, είχαμε εντυπωσιακή αύξηση σε αυτού του είδους την απασχόληση. Κάποιοι δηλαδή δέχτηκαν μερική απασχόληση, ενώ θα προτιμούσαν την πλήρη απασχόληση. Αυτό πάντως δεν μπορεί να είναι η πιο βασική μεταβλητή, άρα θα πρέπει να βλέπουμε τι είδους ε, απασχόληση έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε αυτοί που έχουν μερικές προσφορές να θέλουν, ε, στις περισσότερες χώρες αυξήθηκαν, σε κάποιες χώρες δεν αυξήθηκαν ε, πάνω από 10 μονάδες. Και ο κίνδυνος είναι από 13% στην Τσεχία και σχεδόν 80% στην Ρουμανία, αν κάποιος είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή μερική απασχόληση χωρίς να το επιθυμεί. Ο διάρκειθμός των προσώπων που είναι σε αυτή την κατηγορία στη Ρουμανία διπλασιάστηκε, ή, συγγνώμη, είναι, έχει ποσοστό κινδύνου διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ένωσης. Τώρα, προσωρινά απασχολούμενοι, βλέπουμε εδώ πάλι αποκλήσεις. Πράγματι, Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση στην Εστονία και την Βουλγαρία. Από την άλλη μεριά όμως στο Λουξεμβούργο, στη Λετωνία και στην Αυστρία βλέπουμε αύξηση. Έρχομαι λοιπόν και τώρα στους αυτοαπασχολούμενους. Όπως είπα και προηγουμένως, για να κατανοήσουμε ε, το πώς οδηγούνται στην φτώχεια οι άνθρωποι αυτοί, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ε, αιτίες είναι πολλαπλές. Από την άλλη μεριά δεν έχουμε απαραίτητα τα σωστά στοιχεία από πλευράς των αυτοαπασχολούμενων. Επομένως πιστεύουμε, κυρίως όταν μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους, ότι καλό είναι να δούμε τα πραγματικά στοιχεία της ηλικής ε, φτώχειας. Υπάρχουν λοιπόν χώρες που έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από ότι ε, άλλες. Ε, η Γερμανία, η Σουηδία και άλλες χώρες οι οποίες έχουν γενικά πολύ χαμηλό ποσοστό φτωχών εργαζομένων ε, παρόλα αυτά ε, ε, υπάρχουν προβλήματα ε, λίγους, εργαζό, λίγους αυτοαπασχολούμενους με προβλήματα, σοβαρά προβλήματα εισοδημάτων. ενώ ας πούμε στην Ρουμανία, όπου είναι πολύ σημαντικός ο γεωργικός τομέας, άρα και ο υψηλός αριθμός εποχικών εργαζομένων που εντάσσονται και προσμετρώνται ε, στους αυτοαπασχολούμενους. Ε, ε, εκεί τα στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν το γιατί στη Ρουμανία είναι τόσο ψηλός, ψηλό το ποσοστό. Αυτό τι ήταν μια ε, γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης ε, σύμφωνα με τις μορφές εργασίας. Τώρα θα ήθελα να σας πω τι μπορεί να βοηθήσει ε, για να περιοριστεί ή να μειωθεί η φτώχεια σε καθεστώς όμως εργασίας. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες ελάχιστος μισθός, θα επανέλθω σε αυτό, ε, κοινωνικές ε, μεταφορές έτσι ώστε να αυξηθεί το ε, εισόδημα των οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της στόχης και τρίτο κάποια έμεσα μέτρα, δηλαδή εργαλεία τα οποία μπορούν εμέσως να έχουν κάποια επίπτωση ε, ε, ας πούμε μπορεί να σημαίνει επίδομα για τα παιδιά, μπορεί να σημαίνει δωρεάν περίθαλψη για παιδιά ή για μεγάλους, μπορεί να ε, σημαίνει κοινωνική στέγαση, καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσω κατάρτισης και προώθησης, αύξηση δεξιοτήτων κτλ. Από το 17 είχαμε βρει ότι η εστίαση δεν έπρεπε να είναι όσον αφορά, περισσότερο όσον αφορά τα έμεσα μέτρα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ε, υπάρχουν ε, στρατηγικές ε, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω αυτών των εμέσων μέτρων. Νομίζω ότι το δεύτερο σημείο, social transfers, είναι πολύ σημαντικό. Θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι γίνεται καλύτερα κατανοητή η περιπλοκότητα των, της φτώχειας των εργαζομένων. Πρόκειται για ε, μειονεκτήματα ατόμων και νοικοκυριών ε, που ζουν ε, σε τέτοιες δυσκολίες και που μπορεί να είναι σορευτικά και βεβαίως όλες ε, οι ρυθμίσεις, οι θεσμικές ρυθμίσεις μιας χώρας, οι στρατηγικές οι οποίες έχουν ως στόχο την ποιότητα ε, και την διαθεσιμότητα ε, υπηρεσιών μπορεί να βελτιώσουν, να επηρεάσουν την φτώχεια των εργαζομένων. Πρέπει να εστιάσουμε επίσης την προσοχή μας στον ελάχιστο μισθό. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζουμε από τις μελέτες ότι το ποσοστό των ε, ε, νοικοκυριών που λαμβάνει το ελάχιστο εισόδημα ε, έχει τίνει να προστατεύει αρκετά τον μεμονωμένο ενήλικα απέναντι στη φτώχεια, απέναντι στον κίνδυνο φτώχειας, αλλά συχνά δεν μπορεί να υποστηρίξει πάνω από ένα άτομο. Ε, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει λοιπόν η θέσπιση ελαχίστων ε, μισθών που θα είναι αρκετά υψηλή εάν θέλει κανείς πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους και να αποτρέψει την φτώχεια των εργαζομένων. Επίσης, οι περισσότεροι πολύ συχνά ε, δεν ε, σημαίνει ότι επειδή υπάρχει κάποιος με χαμηλό μισθό θα είναι η οικογένεια φτωχή. Ε, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μόνο ένας ο οποίος κερδίζει χρήματα στο σπίτι και αν υπάρχουν παιδιά κτλ. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα με τον ελάχιστο μισθό είναι ότι προ ώρα αφορά μονάχα τους μισθωτούς ανθρώπους που παίρνουν μισθό. Ε, δεν καλύπτει ακόμα τους αυτοαπασχολούμενους ε, και που είναι επίσης μια πολύ συχνή μορφή εργασίας. Εδώ θα πρέπει λίγο να δουλέψουμε. Δεν έχει γίνει ακόμα πολλή δουλειά για τα θέματα αυτά. Επίσης, ε, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων που πολύ συχνά σε πολλές χώρες δεν καλύπτουν όλες τις μορφές εργασίας και επομένως ε, δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους ανθρώπους που θα έπρεπε να καλύπτονται από τα μέτρα αυτά. Ε, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, επομένως θα φτάσω στα συμπεράσματα. Μπορώ να πω λοιπόν τα εξής. Έχουμε δει ανθρώπους με προσωρινά ε, συμβόλαια, συμβάσει εργασίας, ε, με ε, ανθρώπους που δουλεύουν part-time και κυρίως ανθρώπους που δεν θέλουν, είναι υποχρεωμένοι, αναγκασμένοι να δεχτούν μερική απασχόληση. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει σωστή ε, κοινωνική προστασία ανθρώπων που οι συμβάσεις τους δεν είναι τυποποιημένες, δεν είναι στάνταρ, εκφεύγουν από τις ε, συνηθισμένες συνθήκες. Επίσης είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τον ε, μεγάλη, τη μεγάλη επίπτωση που μπορεί να έχει η γενικότερη κατάσταση του νοικοκυριού ε, στην ε, φτώχεια των εργαζομένων. Επίσης, πιστεύουμε ότι η στρατηγική, η πολιτική θα πρέπει να αναφέρεται σε minimum house income, δηλαδή ε, για το συνολικό εισόδημα το οποίο προκύπτει από το μισθό και από ε, οποιοδήποτε κοινωνικά επιδόματα. Τέλος, θα πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει η φτώχεια και επίσης ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς μετράει αυτή η μέτρηση, μετράει τη σχετική φτώχεια. Ε, και το, τα, την ηλική ε, φτώχεια. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, και οι προτάσεις της Κομισιόν, οι συστάσεις του 2013. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα των παιδιών. Ε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε παιδιά να μεγαλώνουν σε συνθήκες τέτοιας δυσκολίας υπάρχει μεγάλη διασύνδεση ανάμεσα στο, ε, στην οικογένεια με παιδιά, ένα νοικοκυριό με παιδιά και ε, την, ε, τον, τον οικονομικό τους περιορισμό. Η προστασία των παιδιών από τη φτώχεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ο κοινωνικός πυλώνας μπορεί να αποτελέσει ένα καλό στοιχείο ε, το οποίο θα μας οδηγήσει παραπέρα, πιο πέρα από την αρχή των δίκαιων μισθών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας χειροκροτάμε. Ήρθατε από το Δουβλίνο, πολύ δρόμο κάνατε για να έρθετε. Δίνω τώρα το λόγο στους ευρωβουλευτές. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ζητήσετε το λόγο εάν θέλετε να μπείτε στον κατάλογο των ομιλητών να ξεκινήσουμε από τους συντονιστές. Εάν θέλετε το λόγο μπορείτε να το πάρετε, εάν όχι μπορούμε να προχωρήσουμε στους επόμενους ομιλητές. Σε βλέπω ότι και αντιπρόεδρος ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας, για τις αναλυτικές πληροφορίες που μας δώσατε. Δύο ερωτήσεις έχω Είδατε καλές πρακτικές, πολλά υποσχόμενες πρακτικές σε κάποια από τα κράτη-μέλη που να μπορεί να υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε Δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να μας πείτε κάτι. Το αναφέρατε ήδη λίγο, αλλά σχετικά με την πτυχή των δύο φίλων. Και είδατε ε, τι σχέση έχει αυτό με την φτώχεια των εργαζομένων. Αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ντένις, ε, θέλεις να πάρεις το λόγο. Όχι. Ωραία. Από τους σοσιαλιστές. Αγχέλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Δύο ερωτήσεις έχω. Την σχέση ανάμεσα στο ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάτε για τη στέγαση, διότι βλέπω ότι η στέγαση ακριβένει στην Ευρώπη και είδα τα ε, στοιχεία για το Λουξεμβούργο, που είναι πολύ ε, ψηλός ο βασικός μισθός. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει φτώχεια των εργαζομένων. Υπάρχει, υπάρχουν λοιπόν στοιχεία για το ποσοστό που δαπανάτε για τη στέγαση και επίσης έχετε αναλύσει την κατάσταση όσον αφορά τους φόρους που πληρώνουν οι άνθρωποι. Πώς μπορεί η φορολογική πολιτική να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της στόχια των εργαζομένων. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Από το ID κανείς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και κατόπιν το renew, Πρώτα το ID. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γαλλικά. Ίσως να το είπατε αλλά δεν το κατάλαβα. Ποιο είναι το τμήμα, το ποσοστό των εργαζομένων, των φτωχών εργαζομένων ε, εντός των αυτοαπασχολούμενων και κυρίως των εργαζόμενων σε πλατφόρμες. Έχετε κάποια στοιχεία ε, ε, για τα ποσοστά αυτού του συγκεκριμένου κομματιού. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζη. Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Λίτσι. Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της ε, σχέσης ε, ε, που μπορεί να υπάρχει ε, ε, με τους ανθρώπους με αναπηρίες που δυσκολεύονται ενδεχομένω να βρουν και δουλειά και έχουν ίσως χαμηλότερους μισθούς και αν υπάρχει κάποια συσχέτιση. Ευχαριστώ. Την ΚΟΕ. Ο Σλάντε Μερέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και τα πολλά στοιχεία και δεδομένα που μας δώσατε. Καταρχάς, σε μία μικρή παρατήρηση. Μια διευκρίνηση ήθελα να κάνω σχετικά με το γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι φτωχοί ή απειλούνται από φτώχεια ενώ εργάζονται συνήθως ε, με μερική απασχόληση, ενίοτε και σε θέσεις πλήρης απασχόλησης. Αυτό είναι σκάνδαλο όταν μιλάμε για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την ε, ευημερία που επικρατεί εδώ. και βλέπουμε ε, τα τελευταία 10-20 χρόνια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται χωρίς ε, να μπορούν να ζήσουν ε, με το εισόδημά τους. Γνωρίζουμε ότι πιο πολύ επηρεάζονται οι γυναίκες από την κατάσταση αυτή. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι θέλετε να πάρετε το, ως βάση το οικογενειακό εισόδημα, αλλά αυτό στρεβλώνει τα στοιχεία, διότι Κάποιοι άνθρωποι που όσο εργάζονται δεν βγάζουν πολλά χρήματα έχουν μετά και ε, πολύ χαμηλή σύνταξη. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να εξοραίζουμε την κατάσταση και να λέμε ότι είναι το δεύτερο εισόδημα της οικογένειας. Επίσης, ε, μιλήσατε για διάφορες ε, μη τυπικές μορφές εργασίας, την, τους ιονοί αυτοαπασχολούμενους κλπ τι άλλες ε, ομάδες ε, τέτοιων μη τυπικών μορφών εργασίας υπάρχουν ε, που πιστεύουμε ότι είναι ομάδες που απειλούνται περισσότερο από την φτώχεια υπεργολάβους, ιονί απασχολούμενος κλπ. Αυτό θα με ενδιέφερε και θα ήθελα να αναφερθώ και στην εσωτερική αγορά. Έχει επηρεάσει, έχει συμβάλει σε αυτήν την αρνητική εξέλιξη σε κάποια κρατημέλη. Εγώ από τη Γερμανία έρχομαι, αρχές της χιλιετίας, αρχές του αιώνα, Μιλούσαμε για την, ε, τον ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έτσι υπονομεύθηκαν τα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση. Τρία στοιχεία αναφέρατε, το βασικό εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα. Ε, σύντομα θα συζητηθεί αυτό μάλλον και, στην, ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ε, σχετικές προθέσεις. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε το κατόφλι του 60% του ε, μέσου εισοδήματος. Ε, έχετε θέση σχετικά με αυτό και επίσης υπόθηκε ότι θα πρέπει να μιλάμε για έμεσα μέτρα και για τρόπους ανακατονομής του εισοδήματος. Είμαι υπέρ κάτι τέτοιου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Πώς οι άνθρωποι στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη εργάζονται ε, εκτός κάποιο σύστημα συλλογικής ε, σύμβασης ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι απειλούνται από την παγίδα της στόχιας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο από πολιτικές ομάδες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χόμς Καλά το είπα. Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου. Θα προσπαθήσω να, να ε, μάθω καλά, να το, να, το προφέρω καλά μέχρι την επόμενη φορά. Ξέρετε τώρα, Στεχόφσκι λέγομαι και εγώ, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε την Eurofound ε, για την έκθεση που παρουσίασε χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης προσπαθούμε να, δούμε, να βρούμε τρόπο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ποιοτικέ, ε, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και η Ευρώπη αλλά μέσα σε όρους ε, κοινωνικής ε, προστασίας. Ε, η ε, βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν είναι ίδια για όλους. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά την ενεργία, όσον αφορά παιδική ένδυα, όσον αφορά ε, τα κοινωνικά δικαιώματα κτλ. και μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι η πρόληψη της φτώχειας θα πρέπει να αποτελέσει ένα μέρος του γενικού στόχου της μείωσης της φτώχειας. Ε, ένας στους δέκα εργαζόμενους στην Ευρώπη αντιμετωπίζει το φάσμα της ε, φτώχειας και δεν εφαρμόζονται ούτε και οι εγγυήσει για τα παιδιά ε, έτσι, έτσι όπως είχαν συσταθεί από την Επιτροπή. Επίσης, ε, τα, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, των ατόμων δεν αρκούν μερικές φορές έτσι ώστε να αποφευχθεί εντελώς ο κίνδυνος ε, της φτώχειας. Επομένως, πώς βλέπετε ως Eurofund ε, τα θέματα της ε, ευελιξίας στη δουλειά, ε, στην απασχόληση και μήπως θα πρέπει θέματα όπως είναι η κοινωνική ασφάλεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία των παιδιών να τα δούμε με πιο εγκάρσιο τρόπο. και εμείς ευχαριστούμε. Μην μιλάτε πάρα πολύ για να μεταφραστείτε καλύτερα, γιατί δεν πιεζόμαστε από το χρονικό πλαίσιο. Και τώρα ήθελε η κυρία ή ο κύριο Μπίσοπ το λόγο, αλλά αντί αυτού του συναδέλφου θέλει το λόγο κύριο Ντάνιελσον. Ναι, ναι, ναι, θα τα πω πολύ αργά και ευχαριστούμε για τα όσα μας παρουσιάσατε, αλλά ιδίω όσον αφορά τους μη παραδοσιακούς ε, τύπους εργασίας. Και σας ακούσαμε και κανείς δεν θα έλεγε βέβαια ότι θέλει να υπάρχει αυτό το φαινόμενο, όμως εσείς ε, βλέπετε διαφορετικές μορφές από ό,τι τα τελευταία χρόνια κάναμε ε, για τις ε, διάφορες μορφές εργασίας. Ας πούμε, μιλούμε για αυτούς που έχουν παρτική απασχόληση, ε, ε, αυτών που δεν θέλουν να έχουν και στη Σουηδία προσπαθούμε να δούμε πώς ε, να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα δουλεύουν σε πλήρη απασχόληση αν είναι δυνατόν. Από την άλλη μεριά κυρίως έχουμε κάποιες γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στο δημόσιο με τέτοια σχέση εργασίας Οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι φταίει η πολιτική και η πολιτική. Είναι κάτι σαν σύγχρονη μορφή απασχόλησης. Βέβαια, δηλαδή κάποιος στην πράξη έχει δουλειά. Αλλά μπορεί να έχουν διαφορετικού τύπου ε, προσωρινή ε, σύμβαση εργασία και αυτό είναι θέμα που το φροντίζουμε. Άρα υπάρχει στενή σχέση μεταξύ αυτών των μορφών, μη παραδοσιακών μορφών εργασία και τη φτώχεια αυτή. Μα τότε ε, έχουμε το θέμα κάποιων ευρωπαϊκών πολιτικών που πρέπει να γίνουν για να φρενάρουμε αυτό το φαινόμενο. Και πέστε μας, τι θα κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι να έχουν ε, κλασικές μορφές απασχόλησης όπως την πλήρη απασχόληση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάποιος άλλο θέλει κάτι να ρωτήσει, να σχολιάσει. Μπισλάριο. Ευχαριστώ για την εισήγησή σας, τον κύριο Πισλάρο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη διαφάνεια που αφορούσε τις λύσεις. Βεβαίω. Και το λογικό είναι κανείς να προσπαθεί να βρει τις πιο κλασικές σημερινές λύσεις σε σχέση με, δηλαδή, με το ελαχιστή αμοιβή όσον αφορά ε, τις ε, εξαιρετικού χαρακτήρα συμβάσης εργασίας. Τι γίνεται όμως με την διαβιού μάθηση, διάφορες ε, ε, ευκαιρίες που δίνονται για βελτίωση των πραγμάτων όπως κάποιο τους αναβάθμιση. Μας είπατε για αυτή την μελέτη και σε σχέση με αυτά που είπε κάποιος συνάδελφος για πολιτικές και λύσεις. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική που να βελτιώσει τα πράγματα. Ευχαριστούμε. Τελευταίος αλλά ο Μπίσοπ, ο συνάδελφος, ή συνάδελφος Μπίσοπ, συγγνώμη. Μπίσκοφ, Μπίσκοφ μάλλον. Ε, κάτι σε σχέση με αυτές τις ε, ε, προτάσεις μας, δηλαδή ότι έχουμε αντιφατικές πολιτικές στην Ένωση. Δηλαδή, έχουμε αυτές τις συστάσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. πολλέ φορές αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου και οδηγούμαστε σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε για την φτώχεια. Και να άλλη μεριά έχουμε την πολιτική κοινωνία πρόνοια. Πώ μπορούμε να έχουμε κάποια ισορροπημένη αντιμετώπιση μεταξύ της πολιτικής διατηρητικά ταμεία και των οικονομικών μας πολιτικών και έτσι να καταπονημήσουμε το φαινόμενο. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε, Συναδέλφες Κύριε Άρεντ, έχετε το λόγο για 14 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε πολλές από αυτές τις σημαντικές και εύστοχες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στη σειρά που τέθηκαν. Κάποιες ερωτήσεις αλληλοεπικαλύπτονταν κιόλας υποσχέσει ε, σχετικά με εφαρμογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι το ε, ισχυρό σημείο του Eurofound είναι ότι βλέπουμε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες και ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί σε κάποιες χώρες βλέπουμε χαμηλότερα ποσοστά φτώχεια των εργαζομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να ομολογήσω ότι η φτώχεια των εργαζομένων είναι τόσο ε, ειδικό και πολύπλοκο ζήτημα, ε, διότι συνδέεται με ε, το, το, τις θεσμικές ρυθμίσεις και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να κάνουμε γενικεύσεις. Η κρίση στη στέγαση αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα μέτρου που μπορεί να αντιμετωπιστεί διασφαλίζοντας επαρκή και οικονομική στέγη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι ακόμη και σε κάποιες από τις πιο πλούσιες χώρες, αναφέρθηκε το Λουξεμβούργο, Το υψηλό κόστος διαβίωσης σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πάνω από το 1 τέταρτο του εισοδήματός τους δαπανάται για την κατοικία. Αυτή είναι όμως μια πολύ γενική λύση. Γνωρίζουμε επίσης ότι βοηθάει να διασφαλίσουμε οι άνθρωποι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Γνωρίζουμε ότι η φτώχεια των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υψηλή στους ανειδίκευτους εργαζομένους σε χώρες όπως είναι η Ρουμανία ή η Βουλγαρία, όπου υπάρχει γενική έλλειψη στον τομέα αυτών. Ε, θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις ε, ως προς αυτό, αλλά... Ε, υπάρχουν κάποιες λύσεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, αλλά ο Eurofound μπορεί, να συμβάλλει δίνοντάς σας στοιχεία για να δείτε τι κάνουν οι διάφορες χώρες και να συνοψίσουμε την κατάσταση. Αρκετά πολύπλοκο, όπως είπα, κατά τη διάρκεια της ε, παρουσίασής μου είναι το θέμα και θα πρέπει να εξετάσουμε τη σύνθεση των οικοκυριών και να εξετάσουμε ποιο είναι το ελάχιστο εισόδημα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να μην κινδυνεύει από φτώχεια. Γνωρίζουμε ότι πιο πολύ κινδυνεύουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα επειδή οι γυναίκες ε, μάλλον επειδή οι ε, ε, μονογονεακές οικογένειες είναι οικογένειες με μητέρες μόνο συνήθως. Και εάν δούμε τα ποσοστά ανδρών και γυναικών, ε, μπορεί να μην φαίνεται ότι τα πάνε πολύ άσχημα οι γυναίκες, ε, διότι εάν ζουν σε ένα οικοκυριό και φέρνουν ε, σπίτι τον δεύτερο μισθό, μπορεί να είναι δύσκολο να εξηγήσουμε την κατάσταση, αλλά ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας το φύλλο, την πτυχή αυτή. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση τέθηκε σχετικά με το ποιοι είναι οι φτωχοί και για τι πράγμα μιλάμε εδώ. Προσπαθούμε λοιπόν να αναλύσουμε τον εργαζόμενο πληθυσμό σε διάφορες ομάδες και διαπιστώνουμε ότι οι εργαζομένοι σε πλήρη απασχόληση κινδυνεύουν λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με την ε, εντατικότητα της εργασίας. Όσο περισσότερο εργάζεται κανείς, τόσο λιγότερο κινδυνεύει από τη φτώχεια. Όταν φτάνει κανείς σε ηλικία συνταξιοδότηση, ε, αλλάζει η κατάσταση. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλούς φτωχού συνταξιούχους, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που καλύψαμε στη δική μας έκθεση, είναι όμως κάτι που εξετάζει ο Eurofound, ε, τον κίνδυνο της στόχιας ε, μετά τη συνταξιοδότηση. Και εδώ παίζει τεράστιο ρόλο η πτυχή των φύλων. Ε, λόγω του μειονεκτήματος που έχουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ε, δεν κατάλαβα κατά την ερώτηση σχετικά με την περισσότερη φυσιολογική απασχόληση. Τι είδους λύσεις θα μπορούσαν να δοθούν. Νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει περισσότερη δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή, το ερώτημα είναι μάλλον ότι ο καθένας έχει το ίδιο δικαίωμα στην κοινωνική προστασία. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν αν ε, ε, βρίσκεται κανείς σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή αν εργάζεται περιστασιακά ή αν ε, έχει πολλές δουλειές θα πρέπει να έχει κανείς ε, την ίδια κοινωνική προστασία άσχετα από το καθεστώς απασχόλησής του. Πώς μπορούμε να πετύχουμε να εργάζονται περισσότεροι. Αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο. Όσοι εργάζονται βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να τους δώσουμε δουλειά είναι να έχουν πρόσβαση σε καλές, σε ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κατάρτιση καθ' όλη τη ε, διάρκεια της ε, σταδιοδρομίας τους ε, και να έχουν ευκαιρίες προαγωγής. Τα φορολογικά συστήματα συνδέονται με την κοινωνική ανακατανομή του χρήματος. Θα πρέπει λοιπόν να δίνονται φορολογικές, να δίνεται φορολογική ανακούφιση ε, σε, στους φτωχούς, ε, αλλά και αυτό εξαρτάται από την κατάσταση στην κάθε χώρα. Εμείς ε, μπορούμε να προσφέρουμε το εξής, να καταγράψουμε τις ερωτήσεις αυτές και να υποβάλλουμε προτάσεις ε, αντί να προσπαθήσω τώρα ε, να σας ε, ξεπετάξω στα γρήγορα κάποιες ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να συζητήσουμε πολύ περισσότερο εις βάθος το θέμα αυτό, διότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Έχουμε κάποιους πρώην πρωθυπουργούς, πρώην ε, ε, υπουργούς απασχόλησης ε, που έχουν πολλές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά και για τον ελάχιστο μισθό. Ελπίζω σε κάποιες μελλοντικέ συζητήσεις ε, να μας απασχολήσει επίσης το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Also, now I will... Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, που είναι η γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης για τη θέσπιση του προγράμματος διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Ο κύριος Δράγος Πίσλαρου από το Ρινιού είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Και θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή για να σχολιάσει το, το σχέδιο γνωμοδότησής του. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεύτερο θέμα σημαντικού ενδιαφέροντος. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο προέκυψε από την ανάγκη να προσέξουμε περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις μας ε, ε, που προωθούμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν οι συστάσεις αναχώρα που υποβάλλονται ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά μόνο το 1 τρίτο εξ αυτών γίνεται σεβαστό στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που ε, σχεδιάζονται οι μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από το Μάιο του 2018, ε, είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που στόχο έχει να βοηθηθούν ε, οι χώρες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Συγκεντρωνόμαστε στην σημασία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων παρέχοντας κίνητρα και προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο σκοπό η κατάσταση προφανώς ε, μας κάνει να θέσουμε το ερώτημα γιατί έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ τα πράγματα. Όλα ξεκίνησαν ε, πάλι το 2018, υπήρξαν κάποιες πρώτες συζητήσεις όπως βλέπετε στην ε, διαφάνεια και τον Δεκέμβριο του 2018 είχαμε διάσκεψη κορυφής που ενέκρινε το αρχικό πλαίσιο αυτού του ε, δημοσιονομικού μέσου που λέγεται BIC ε, για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Τον ε, Φεβρουάριο είχαμε σχέδιο έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2019 σχετικό έγγραφο. Κατόπιν είχαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ λάβαμε από τη Φιλανδική Προεδρία μια κάπως διαφορετική εκδοχή του εγγράφου και από εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω για να καταλάβετε όλοι τι συζητάμε εδώ. Όπως λοιπόν βλέπετε στη διαφάνεια, η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερόταν στο εργαλείο για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που ε, κάλυπτε την ε, ζώνη του ευρώ και τις άλλες χώρες ε, με αντίστοιχα 17 δισεκατομμύρια 5 δις. Κατόπιν έχουμε και το στοιχείο για την διευκόλυνση για τη σύγκληση και την τεχνική υποστήριξη. Από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με βάση τις συζητήσεις στην ε, διάσκεψη υψηλού επίπεδου και στο ΕΚΟΦΗΝ στο Συμβούλιο, προέκυψε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο με τρία διαφορετικά μέσα. Από τη μία λοιπόν έχουμε το BIC, το Δημοσιονομικό Εργαλείο για τη Σύγκληση και την Ανταγωνιστικότητα, το οποίο αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται, αλλά προσέξτε τώρα, ε, επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για χώρες της Ευρωζώνης ε, και ε, τα άλλα κράτη-μέλη. Κατόπιν έχουμε ένα δεύτερο εργαλείο για κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη που λέγεται ε, μέσω σύγκλησης και μεταρρυθμίσεων, ε, λέγεται κρί δηλαδή, είναι το ακρονίμιο, και κατόπιν έχουμε την τεχνική υποστήριξη που παραμένει λίγο πολύ είχε. Τι είναι σημαντικό εδώ λοιπόν και γιατί σας κάνω αυτή την εισαγωγή, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια γνωμοδότηση πάνω στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ Η κατάσταση καθορίζεται από το τελευταίο έγγραφο της Φιλανδικής Προεδρίας. Τούτου λεχθέντος, κατά τη σύνταξη της νομοδότησης, κάνουμε το εξής. Στις 13 ε, Ιανουαρίου παρουσίασαμε τα διάφορα στοιχεία ε, εντός ε, του χρονοδιαγράμματος. Είχαμε τις μεταφράσεις μέχρι τις 24 Ιανουαρίου και με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υπάρχει προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 19 Φεβρουαρίου. Δεν απομένει λοιπόν πολύς χρόνος και πάλι όμως το έγγραφο αυτό είχε υποβληθεί ήδη στις 24, ήταν διαθέσιμο το έγγραφο στις 24 Ιανουαρίου. Υποτίθεται λοιπόν τώρα ότι το Μάρτιο θα πρέπει να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες, ε, να εκπονήσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες ε, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και προβλέπεται στις 29 Απριλίου η ψηφοφορία στην ΕΜΠΛ και στην Νίκον και στην Μπάτζ 27 και 28. Συνάδελφοι, λοιπόν, ε, όσον αφορά το περιεχόμενο, εγώ προτείνω 24 τροπολογίες, 13 ε, για τις αιτιολογικές σκέψεις ε, και 11 για τα άρθρα και θα αναφερθώ στα βασικά στοιχεία που τροποποιούμε. Καταρχάς, το πνεύμα της Επιτροπής ΕΜΠΛ ε, ε, παραπέμπουμε στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την απασχόληση, την προσβασιμότητα της υπηρεσίες για την απασχόληση αλλά και για την νεολαία. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για την Επιτροπή Απασχόλησης. Όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο και να τονίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και η κοινωνική Ευρώπη, όπω παρουσιάστηκε από την πρόεδρε τη Επιτροπή Ursula von der Leyen και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνδεθούν με το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε επιτάπητο. Ε, κάτι πολύ σημαντικό που προτείνουμε επίση είναι ότι οι μεταρρυθμίσει δεν θα πρέπει να γίνουν κατανοητέ ε, μόνο ε, σε σχέση με την κρίση, τα μέτρα λιτότητας που οδηγούν στη φτώχεια. Πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις για να γίνει κατανοητό το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να είναι μεταρρυθμίσει που ε, ε, επιτρέπουν την προσβασιμότητα και που δημιουργούν ευκαιρίες. Και θα θέλαμε να τονίσουμε, και γι' αυτό έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία, ότι ιδιαίτερα οι ευάλωτε ομάδες ε, θα πρέπει να στοχεύονται όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και την ε, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Χρειάζεται τεχνολογική ανάπτυξη, χρειάζονται θεκτικές αγορές εργασίας και αυτό σχετίζεται με το θέμα που συζητήσαμε πριν. Σχετίζεται με τις νέες μορφές απασχόλησης, την εργασία σε πλατφόρμες και όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη φτώχεια και την απασχόληση. Κάτι ακόμη που προτείνουμε σε τροπολογία σχετίζεται με τις ε, μη ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για σύγκληση. Η ε, προσχώρηση στο ευρώ ε, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε μεταρρυθμίσεις που να προωθούν τη σύγκληση και όπου έχουμε σημαντική ε, σύγκληση. Και μάλλον ε, προτείνουμε τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να υπάρξει η σύγκληση. Ε, είναι πολύ σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις χωρίς αποκλεισμούς για την κοινωνική σύγκληση. Και θέλουμε να τονίσουμε την σημασία της υποστήριξης που προβλέπεται από τα θεσμικά όργανα και όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη. Επίσης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την επιλεξιμότητα των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην παρούσα σύνοδο του Κοινοβουλίου συζητάμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σημαντικό είναι να τονίσουμε τους κοινωνικούς δείκτες στα κράτη-μέλη. Και τέλος, αλεξίσου σημαντικό, ε, θέλω να αναφέρω την ενθάρρυνση των κρατών μελών ε, που ε, θέλουν να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά, να έχουν διαβουλεύσεις με ομάδες ενδιαφερομένων, με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που καλύπτω με τη γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας και πάλι ότι υποβάλαμε τροπολογίες με βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με βάση τις αρχές που έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, σημαντικό είναι ότι στις 17 του μήνα έχουμε το Eurogroup, στις 20 έχουμε την ECOFIN και με βάση αυτά θα έχουμε την τελική εκδοχή του ε, κειμένου στο οποίο βασιζόμαστε. Έτσι λοιπόν υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό, διότι ακολουθούμε εδώ μια διαδικασία η οποία σε κάποιο βαθμό μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Τούτου λεχθέντος και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας παρουσιάσω την νομοδότησή μου. Το πιο σημαντικό στοιχείο της συζήτησης θα είναι φυσικά οι ερωτήσεις και πολύ θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Είμαι και συνεισηγητής ε, εκ μέρους του Κοινοβουλίου για το συνολικό θέμα. Θα είναι λοιπόν πολύ καλός αυτός ο τρόπος να μεταφέρουμε τις θέσεις της ΕΜΠΛ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank your... Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, όχι, όχι, όχι, διορθώνει η γραμματεύσα πρώτος πρώτος θα αγορεύσει η συνάδελφος Κλάρα, γιατί ο Χωσιμον Φερνάντες δεν παρίσταται, οπότε Κλάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ να σας τα πω σύντομα πρώτα πρώτα, λέει η κυρία Ντόμπερτ. Καταρχήν, όλοι νιώθουμε κάποια απογοήτευση από την ε, πρόταση γενικώς όπως το είπαμε εδώ και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει αυτό κάπως να το εκφράσουμε και τους προβληματισμούς μας και την ανησυχία μας. Τώρα συγκεκριμένα όσον αφορά για το πρόγραμμα της μεταρρύθμισης, μου αρέσει η προσέγγιση του εισηγητού και θα ήθελα να σας τονίσω τρία τεινά που νομίζω ότι έχουν σημασία. Και επίσης να υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες Οπότε να είμαστε όσο γίνεται για τα τρία ε, θέματα που μας απασχολούν πιο συγκεκριμένοι γιατί είναι σημαντικό. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καλύψουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και θα πρέπει να ε, θωρακίσουμε την κοινωνική διάσταση γενικώ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το έργο μας αμέσω επόμενους μήνες, μήνες ή χρόνια σε σχέση με τις διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίω ότι έχει σχέση με το MFF, το πολιτισμό με πλαίσιο ή τον προπολογισμό. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την διαβούλευση με κοινωνικού εταίρου, ακριβώ όπω τα ε, τόνισε ο Θα πρέπει αυτό να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο και να μπορέσει η Επιτροπή να ασκήσει κάποιο είδου ε, ε, διασταύρωση. Να μην βάζει απλώ φραγίδα και υπογραφή. Θα πρέπει να βλέπει τι ισχύει στην πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή η διαβούλευση ε, τους γενικούς εταίρους, όλα αυτά με την εμπειρία τόσων ετών. Δεν γίνονται αλλιώ εκεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. γι' αυτό και σας λέω θα είναι σημαντικό να γίνει έτσι το πράγμα. Επίσης κάτι άλλο. Σέντεβο. Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μόνο το μέγεθο του πληθυσμού για την διάθεση των κονδυλίων. Το θέμα μας εδώ είναι η ελεγγύη και η συνοχή. Αυτά έχουν σημασία για την κοινωνική πρόνοια, τον κοινωνικό πυλώνα. Οπότε εγώ θα υποβάλω μέχρι την πέμπτη της τροπολογίες μου για αυτά που σας ανέφερα. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ελαφρώς εκτός θέματος ότι βέβαια το πρόγραμμα υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων έχει την εξή λογική. Το κράτο μέλο θα πρέπει να το ζητήσει. Αλλά για τα συγκεκριμένα προγράμματα και έργα και χρηματοδοτικά προγράμματα Έχουμε τι οργανώσει τι κοινωνικέ, των πολιτών κλπ. Όλοι αυτοί που καλύπτονται από το πρόγραμμα, που εμπλέκονται και άρα θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι θέματα αντιμετωπίζει η κάθε χώρα. Αυτό να κάνουμε στο εξάμεινο που προβλέπετε, διότι ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποια με πρόοδο, αλλά για λόγους πολιτικούς τα κράτη-μέλη μπορεί να μην θέλουν να κάνουν τα παρακάτω βήματα που απαιτούνται ε, επίσης οι τοπικές περιφερειακές αρχές, ε, έρευνες, ε, δημοσιεύσεις, μελέτες, ούτως ώστε να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα, γιατί αυτό χρειάζεται για την ευάδειση της Ένωσης κλπ. Προβλέπονται κονδύλια για τα κράτη-μέλη, δεν θα φύγουν Έχουμε και τις ε, συγκεκριμένες ειδικέ συστάσεις, τις εκθέσεις κάθε χώρας κλπ. Αυτά θα προτείνω με τις τροπολογίες μου. Επίσης, πολύ σχετικό είναι το θέμα του μέσου διευκόλυνσης της σύγκλησης. Υποχρέωση εισόδου στην Ευρωζώνη. Εάν δεσμεύτηκαν να το κάνουν. Και θα δούνε τα καλά του ευρώ. Όμως Κάποια κρατημέλη για πολιτικούς λόγους δεν θέλουν και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, εάν αυτό είναι δέσμευση νομική των κρατών μελών, ε, τότε θα πρέπει και άλλοι να βοηθήσουν με μελέτες, με καμπάνιες και έτσι να συγχθεί αυτή η κοινή προσπάθεια προς το ευρώ ως βάση για την οικονομία. Τώρα, τελευταίο. Η γενική προσέγγιση ε, προβλέπει την προχρηματοδότηση και έχουμε όλα αυτά που σας είπα και ξέρω ότι τώρα άλλα λέμε, δεν είναι αυτό το θέμα προχρηματοδότηση προγραμμάτων, αλλά θα πρέπει σε κάποια προγράμματα η προχρηματοδότηση να προσεχθεί ιδιαίτερος, να δούμε τι θα προβλέπετε αν θέλουμε να υπάρχει εμπλοκή και να βοηθήσουμε τοπικές αρχές και φορείς των πολιτών. Νομίζω πως πρέπει να κινηθούμε έτσι. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε Κλάρα. Έλενα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε αυτή την πρόταση για τον κανονισμό που αποτελεί ένα μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την συμβολή ε, για τα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά τις διευθυντικές αλλαγές προβλέπει η Επιτροπή. Εγώ νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολες κάποιες ε, εφαρμογές αποφάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεσμεύονται τα κράτη-μέλη. Πρέπει να εκτελέσουν τις αποφάσεις της Ένωσης όσον αφορά την οικονομική πολιτική, την κοινωνική πολιτική και ό,τι τυχόν προκύψει. Ε, πρόκειται για πολύ σημαντικά ε, συνέπειες. Στην Ιταλία ακόμα πληρώνουμε την ύφη για τις μεταρρυθμίσεις της Κομισιόν. 11-12 μεταρρύθμιση Φορνέρο επί Μόντι και την εργασιακή νομοθεσία του 11 της κυβέρνησης Ρέντσι. Όταν έγινε η εισήγηση της Κομισιόν αναφέρθηκε η τεχνική αρρωγή για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προς ε, την Ελλάδα από την Κομισιόν και την Task Force 11 ε, με 13 αλλά βγήκε κάποιο είδους αξιολόγηση θετική για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα εκείνων των μεταρρυθμίσεων. Επομένως, θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνοχή, καλύτερη παραγωγικότητα, απασχόληση, κίνητρα επενδύσεων, βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε έχουμε το πράγμα της Ιταλίας. Ε, εκεί επιβλήθηκαν απολύσεις, ε, αναστάτωση στην απασχόληση. Τι να πω για την ε, Ελλάδα. Τα ξέρετε από τις εφημερίδες. Τα ανάποδα, τα αντίθετα γίνανε. Οπότε εμείς ως ομάδα δεν θέλουμε οι Βρυξέλλες να υπαγορεύουν τις μεταρρυθμίσεις Πού είναι η εθνική κυριαρχία. Είμαστε κάθετα εναντίον για αυτό το πρόγραμμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης. Και η αρμοδιότητα για φορολογικά, νομισματικά θα πρέπει να είναι εθνική. Για επενδύσεις, κατάλληλο πώληση μίξ κλπ.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 ε, αγαπητέ συνάδελφε Πισλάροφ, ε, για το φιλόδοξο αυτό ε, πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά αφορά ένα σημαντικό πρόγραμμα και που σχετίζεται βεβαίως και με τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό. Τα υπόροι οι οποίοι αφορούν το πρόγραμμα 21-27 και αποτελείται από 25 ευρώ και τον ε, καταμερισμό τους, για την βελτίωση της ε, ε, κοινωνικής κατάστασης, του περιβάλλον κτλ. Η κατανομή αυτή οπωσδήποτε θα βελτιώσει τις συνθήκες στους τομείς αυτούς και επομένως μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα αναφέρονται στην γνωμοδότηση. Δηλαδή ότι οι πόροι αυτοί μπορούν να έχουν σημαντική αντίκτυπο στην κοινωνική κατάσταση αλλά και στην, αγορά, την κατάσταση της αγοράς της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ε, μέσα από την κατάρτιση, μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των ικανοτήτων όλων έτσι ώστε όλοι να έχουν ε, περισσότερες ευκαιρίες και επομένως οι νέοι να έχουν ε, καλύτερο μέλλον και εν τέλει να βελτιωθεί και το γενικότερο σύστημα της κοινωνικής προστασίας. Ε, ε, τα συστήματα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία είναι συστήματα τα οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα ε, να αντιμετωπιστούν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξή σε σχέση με την γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συνεκτικοί στο, σχολιασμό, δηλαδή τα σχόλιά μας θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα και οπωσδήποτε θεωρώ ότι σκόπιμο είναι να μην επιμηκυνθεί ιδιαίτερος το έγγραφο αυτό, να μην γίνει δηλαδή ιδιαίτερα μακροσκελές, έχει συζητηθεί επανειλημμένα ε, και ε, προβλέπονται και συγκεκριμένα εργαλεία πλέον στο ιστορικό το Πιστεύω πάντως ότι ορισμένες ε, διατυπώσεις είναι υπερβολικές, δεν βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου, το περιπλέκουν άνευ λόγου και επίσης το κάνουν πολύ πιο μακρύ χωρίς λόγο επίσης. Αλλά και εμείς θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώνα. Δεν βλέπω, λέει ο Πρόεδρος, την κυρία Μαρία Μπέγκρα Χάνσεν ή κάποιον από τους πράσινους. Θα δώσω το λόγο στην Σάντρα Περέιρα από την GUNGL. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εργασία του. Πρόκειται εδώ για θέματα τα οποία είναι ε, σημαντικά και εμείς έχουμε διαφορετικές απόψεις. Το 2018 υπευλήθη, παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή προοπτική. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ούτε οι διαπραγματεύσεις, ούτε αυτή η γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης μας άλλαξαν ε, γνώμη. Στην ουσία αντικατοπτρίζονται οι προτάσεις της ε, ε, Γερμανίας ο στόχος είναι να, να υπαγορευθούν και να υποχρεωθούν στις χώρες και να υποχρεωθούν οι χώρες να ακολουθήσουν αυτές τις ε, τις μεταρρυθμίσεις. Ε, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, όμως, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντιτίθενται στα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς επίσης αντιτίθενται και στις αρχές της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Ε, η κάθε χώρα χρειάζεται διαφορετικά μέτρα και αυτό πρέπει να γίνεται και βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντας ε, ε, υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση ανά χώρα όμως και μέσα από τέτοιου είδους προτάσεις ε, στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμειγνύεται στα εσωτερικά ε, των ε, χωρών και εν τέλει δεν μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εμείς πιστεύουμε ότι αναφορές στους τόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της συνοχής της δημοκρατίας, να συμπεριλαμβάνονται δηλαδή σε αυτήν ε, την γνωμοδότηση στην ουσία θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή τη δημιουργία ενός αντικοινωνικού, αντιεργατικού προγράμματος. Ωραία, θα ζητήσω τώρα από την Κομισιό να μου πει αν θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε, παρακαλώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πλιστάρο για την ε, έκθεσή του, καθώς επίσης και για τις ε, σωστές εξηγήσεις τις οποίες ε, έδωσε. Έγινε μια πρώτη πρόταση από την Κομισιόν και από αυτή τη βάση εργάζεται και το Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα ποιο θα είναι το κείμενο. Έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και θα υπάρξουν και περαιτέρω τροποποιήσεις πιστεύω στο, κείμενο. Ωστόσο ο βασικός στόχος παραμένει ίδιος η υποστήριξη των διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων. Η ιδέα δεν είναι να υπογραμμίσει, συγγνώμη, να ε, ε, υποδεικνύει η Κομισιόν ή να υπαγορεύει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη ε, οτιδήποτε, απλώς πρέπει να διασφαλιστεί ε, η συνέχεια στα κράτη-μέλη και βεβαίως να διασφαλιστεί και η οικονομική υποστήριξη των ε, ε, αρχών. Γι' αυτό λοιπόν ε, έγινε η πρόταση για μια ε, δέσμη τέτοιων μέτρων. Η ιδέα βεβαίως είναι ε, να μπορέσει να υλοποιηθεί η βελτίωση των, και η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε όχι να μειωθούν τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά αντιθέτως να υπάρχουν περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, να καλυφθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτή η κοινωνική ε, διάσταση ε, και ε, να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν την ισότητα έτσι ώστε να προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε μέσω τέτοιων προγραμμάτων να γίνει η κοινωνία και κοινωνικά και οικονομικά πιο ανθεκτική. Επίσης κάποιες τροποποιήσεις ε, στην αρχή προτείνεται εκ των προτέρων εξάντε κλίδα κατανομής στη συζήτηση με το ε, Συμβούλιο. Ε, το Συμβούλιο θέλει και ένα επιπλέον στοιχείο, δηλαδή το ΑΕΠ. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα τμήμα το οποίο δεν έχει αλλάξει καθόλου ε, σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν και μετά από εξέταση ε, του ε, Συμβουλίου. Στην ουσία εδώ θα υπάρξει μια συνέχεια του προγράμματος, του ήδη υφισταμένου προγράμματος της Κομισιόν. Επίσης, τεχνική βοήθεια μπορεί να υπάρξει σε θελοντική ε, βάση από πλευρά της ε, Κομισιόν. Επίση, αξιολόγηση λαμβάνει η χώρα τώρα και σύντομα ε, θα είναι διαθέσιμη. Αυτό θα γίνει λοιπόν και θα έχετε τα αποτελέσματα όσον ούπο. Επίσης, σε αυτά τα πλαίσια η ιδέα είναι ότι οι αρχές θα κάνουν τις ε, προτάσεις και όσον αφορά τις δέσμες και όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη και επομένως Ε, ενδεχομένως τοπικές αρχές θα μπορούσαν να είναι έμεσα ή άμεσα ε, ε, δικαιούχοι. Τα, στην ουσία όμως τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα παίρνουν τις αποφάσεις. Ε. Η Κομισιόν δεν έχει εδώ, δεν μπορεί να ε, ε, εισάγει οποιασδήποτε απαιτήσει, γιατί αυτό θα σήμαινε ανάμειξη στα εσωτερικά Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να δούμε και την ικανότητα ολοκλήρωσης ε, και ε, υλοποίησης από πλευράς των κρατών μελών και οπωσδήποτε σε περίπτωση που μιλάμε για τοπικές περιφερειακές αρχές θα πρέπει η Κομισιόν να είναι βεβαία ότι αυτές οι αρχές έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες. Παραπέρα όμως δεν μπορεί να πάει η Κομισιόν. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και βεβαίως είμαστε ε, στη διάθεση και των δύο ε, ε, εισηγητών για συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας μόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η παρέμβαση που έκανε η Κομισιόν ξεκαθάρισε κάποια στοιχεία, ας πούμε το θέμα των κριτηρίων, ναι, γιατί είναι γεγονός ότι ο, εκτός από τον πληθυσμό έχει προσθεθεί και το κατακεφαλή εισόδημα και το ΑΕΠ εξεπλάγει είναι θετικά Ε, ότι ενδεχομένως ε, μέσω του άρθρου 23 τώρα μπορούν να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ε, και θεσμοθετημένοι οργανισμοί και περιφέρειες κλπ. να χρησιμοποιηθούν λοιπά Μπορεί να είναι τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, μπορεί να είναι κάποιες οργανώσεις εργαζομένων κλπ. Ένα άλλο θέμα, τα CSR και το όλο σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ενδεχομένως ε, μπορεί να μην προκύπτουν οι σωστές συστάσεις γιατί δεν ισχύουν όλα, όλες τις χώρες μέλη. Ωστόσο, αυτά που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο ε, μια και, ε, ε, τείνουν ακριβώς και στο να εμπλέξουν και την κοινωνική, ενδεχομένως ακόμα τώρα και την περιβαλλοντική πτυχή στην, στα πλαίσια του εξαμήνου και ο στόχος είναι η ενίσχυση του εξαμήνου και το εξάμεινο να γίνει πιο ισορροπημένο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα και συνέχεια, συνέπεια ανάμεσα στα, στους διάφορους φακέλους που συζητούν εγώ θεωρώ ότι η Κομισιόν μπορεί να κάνει καλές ε, συστάσεις πρέπει να δουλέψουμε μαζί τους έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο. Ε, η Κομισιόν, και το λέω και το ξαναλέω και μία ακόμα φορά, η Κομισιόν δεν είναι ο εχθρός μας. Μπορεί να είναι και αρρωγός μας. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ε, ε ξαναείπα ότι η διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις στο συλλογικό θυμικό έχουν αρνητικό πρόσημο. Ωστόσο, είμαστε μια κοινωνία η οποία πλέον ε, βασίζεται στις ευκαιρίες και στην πρόσβαση. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ρίτσι, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η ιδέα βεβαίως εδώ είναι στο πρώτο μπίξ, στο πρώτο εργαλείο, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε να μην γίνουν επενδύσεις, να μην γίνουν ε, ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά επενδύσεις και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να απαντήσει στις ανησυχίες σας. Για μία ακόμα φορά λέω ότι τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ δεν, ε, δεν είναι υποχρέωση. Εδώ έχουμε ευκαιρίες, εδώ έχουμε κίνητρα έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις αλλά και σε επενδύσεις. Τέλος, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα σχόλιά σας. Περιμένω ε, τις τροπολογίες και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και μια πολύ καλή συζήτηση έτσι ώστε ε, εν τέλει η Επιτροπή Απασχόλησης, η Επιτροπή μας ΕΜΠΛ ε, να κάνει μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν και θα περιμένουμε και την επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ντράγκος. 19, Φεβρουαρίου του 2020 στις 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε 12 μη ή 12 μη μη, πάντως είναι 12 το μεσημέρι για να, γίνουμε, να το καταλάβουμε όλοι. 29 Απριλίου στην Έπλεθα... ε, συζητηθεί το θέμα και η τελική ψηφοφορία 27 ε, Μαΐου και ε, συζήτηση και ψηφοφορία τελική στην Ολομέλεια, στην Ολομέλεια του μηνός Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την ε, ωραία συζήτηση. Έχουμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή. Τώρα θα μιλήσω όμως τσέχικα. Άρα βάλτε τα ακουστικά σας. Ε, γιατί εγώ θα κάνω κάποια σχόλια από πλευράς Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ε, καλωσορίσω τον κύριο Πρέ Λάρου Τούρου, Γενικό Εισηγητή της Επιτροπής Μπούτζ. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που έχω να πω δύο λόγια σχετικά με τη ε, διαδικασία του προπολογισμού και να σας πω ποιο είναι ο προβληματισμός μου ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, στο παρελθόν είδαμε ότι οι γνωμοδοτήσεις και οι προτεραιότητες των επιτροπών που έκαναν μόνο γνωμοδοτήσεις για τον προϋπολογισμό στην ουσία λίγο επηρέαζαν το, την τελική εκδοχή του προπολογισμού. Χαίρομαι λοιπόν τώρα που και η Επιτροπή Απασχόλησης αλλά και άλλες επιτροπές εμπλέκονται στη διαδικασία περισσότερο από πριν προς ώρας ε, δεν μπορώ να πω εάν η αλλαγή αυτή ε, θα βοηθήσει έτσι ώστε να προωθηθούν κάποιες δικές μας προτεραιότητες στον τελικό προϋπολογισμό. Ωστόσο παραμένω αισιόδοξο γιατί εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί. Θα ήθελα να ευχαριστώ, ευχαριστήσω την Επιτροπή Προϋπολογισμού για την θέση και τη στάση τους. Ε, μια άλλη επιθυμία μου και ευχή μου έχει περισσότερο τυπικό διαδικαστικό χαρακτήρα για την δυνατότητα να επαναεισηγηθεί μια τροπολογία ή ε, στην Ολομέλεια εάν αυτή η τροπολογία έχει απορριφθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Βάσει του 4 του ιστορικού κανονισμού αυτό είναι δυνατό, αλλά είναι μια θεωρητική δυνατότητα, γιατί στην πράξη, στην ουσία σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από μια ε, ιδιαίτερα αντιφατική, αντικρουόμενη τέλο πάντων διαδικασία στην αντίστοιχη επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως ε, ε, Ξέρουμε τι συμβαίνει. Ε, κάθε χρόνο υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες ε, όταν επανεισάγονται, επανυποβάλλονται δεν γίνονται δεκτές, απορρίπτονται και στην ε, Ολομέλεια. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι τα πιλωτικά προγράμματα μόνο θα πρέπει να γίνονται δεκτά αυτά που ε, είναι A ή e B. Αλλά πάντο, δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι πάντοτε αντικειμενική η κρίση της ε, Επιτροπής και οποτεδήποτε βλέπουμε εμείς αυτές τις ελλείψεις θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα είτε στις Επιτροπές είτε στην να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ε, επανυποβολή τροπολογιών. Αλλά το θέμα είναι ε, πώς θα κερδίσουμε χρόνο και χρήμα, πώς θα βελτιώσουμε τη διαδικασία. Ε, δηλαδή ή θα πρέπει ή θα πρέπει να διαγραφεί αυτή η δυνατότητα ε, ή θα πρέπει αυτόματα να προωθούνται ε, τα, οι τροπολογίες αυτές ή τα μέτρα αυτά. Εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είμαι βέβαιος ότι και σε άλλες επιτροπές ε, θα υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα εδώ να σας δραχτώ τη ε, ευκαιρία ε, κύριε Λαρουτουρού που είσαστε εδώ έτσι ώστε να σα πω αυτά που με προβληματίζουν από την άλλη πλευρά βεβαίω. να σα πω ότι ε, τώρα θα σα δώσω το λόγο γιατί γι' αυτό ήρθατε εδώ για να μα μιλήσετε παρακαλώ Ακόμα και για του Γάλλου είναι το όνομα μου δύσκολο να το προφέρει. Σα ευχαριστώ για την φιλοξενία Ευχαριστώ. Από την άλλη μεριά συμπαθάτε με γιατί είμαι μέλος ε, της Επιτροπής ε, Απασχόλησης αλλά είμαι και εισηγητής στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Νέος βουλευτής, είμαι εδώ λίγους μήνες και έχω πάρα πολλή δουλειά. Θα πρέπει να πάω σε όλες τις επιμέρους επιτροπές, στο Βερολίνο επίσης, για να τις κάνω τις σχετικές διαπραγματεύσεις και οπότε συμπαθάτε με γιατί δεν είμαι και τόσο δυναμικό μέλος της Επιτροπής μας. Πάντως εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαι με πασχόληση και καταπολέμηση της φτώχειας. Σήμερα ήρθα όχι να σας παρουσιάσω μόνο τις κατευθύνες γραμμές, αλλά επειδή συμφωνώ με τις ανησυχίες σας, υπάρχει βάσιμος λόγος ανησυχία σε σχέση με το σχέδιο του προπολισμού από το Συμβούλιο. Ο Σολ Μισελ το Φεβρουάριο θα κάνει μια σχετική συνάντηση ε, είναι πολύ αδύνατος 1,074 του ΑΕΠ. Αυτό είναι αστείο ποσό, αστείο ποσοστό. Δεν είναι δυνατόν εμείς να δεχτούμε τέτοιο φτωχό προπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος για κλίμα, κοινωνικά, προσφυγικό, για όλα τα σημαντικά. Και οι προηγουμένες πολιτικές ομάδες ήδη έχουν αντιδράσει αρνητικά, άρα πρέπει να έχουμε ενίο μέτωπο. Γι' αυτό και συναντά όλες τις ε, Επιτροπέ, Είπαμε είμαι ευρωβουλευτή σε 6 μήνε. ε, τη για τον προηγούμενο του 20, 1,9 δι τόσα κερδίσαμε, περισσότερα από όσα ήθελα να δώσει το Συμβούλιο και αυτό, γιατί πέντε πολλοί ομάδες ήταν ενωμένε. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Οπότε αρχίσαμε το Συμβουλίο αυτή την προσπάθεια για να γνωριστούμε. Ε, και να δούμε θα καταλήξουν τα πράγματα και οι διαπραγματεύσει οι δύσκολε τον Φεβρουάριο. Γενικώ ο μόνο εισηγητή για τον προηγούμενο του 21. Κοινό μέτωπο, να δούμε τι γίνεται με το πολιτέ πλαίσιο και πολλά από αυτά που λέω όταν πάω στο χρόνο και αλλού βεβαίω αφορούν και τους διαπραγματευτέ μας Όλοι μαζί προσπαθούμε. Ήρθα εδώ μόνο να ψάξω συμμάχους γιατί θα πρέπει να υπάρχουν σύμμαχοι. Είπαμε οι πέντε ομάδες για να κερδίσουμε την ε, μάχη και αντί να λέμε πράγματα δεξιά και αριστερά θα πρέπει να λέμε κάθε χώρα τι προτεραιότητες έχει συγκεκριμένα παραδείγματα για να πείσουμε τους αγικού κρατών και κυβερνήσεων και να κερδίσουμε τον κόσμο. Επίσης, έχω εδώ πέρα ένα PowerPoint Έχουμε δύο προτεραιότητε επομένως στον προϋπολογισμό του 2021. Κλίμα, απασχόληση και κοινωνική δικαιοσύνη. Για το κλίμα. Είχα πάει στο Μαλί, στο Μπαμάκο και είπαν στο Σαχέλ έχει τώρα μια ξηρασία που δεν έχει προηγούμενο. Ποτέ τόσο άσχημα τα πράγματα το AIDS βέβαια ε, είχε πολλά θύματα, αλλά τώρα θα είναι ακόμα περισσότερα τα θύματα. Είναι κάτι σαν AIDS του κλίματος και έχουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Πήγα και σκέφτηκα ένα παρατηρητήριο που μετράει το διοξείδιο. το φτιάξαν αυτό το μηχάνημα, αυτό το παρατηρητήριο οι Αμερικάνοι και 0,8 μονάδες κάθε χρόνο. Στην αρχή τώρα έχουμε τρεις φορές περισσότερη αύξηση έχουμε πάει στις 4-15 μονάδες και βλέπουμε ότι σε καμία μας χώρα δεν γίνεται τίποτα. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ένας φαύλος κύκλος. Και έχουμε αυτές τις δασοπυργαγίες στην Αυστραλία, δημιούργησαν ε, ε, διοξίδιο, ε, περμαφρόστ λοιπά. Ακόμα χειρότερα. Οπότε είχα πάει στη Μαδρίτη το Δεκέμβριο για στη διάσκεψη για το κλίμα. Ε, όλοι προσβλέπουν στην Ευρώπη και όλοι μαζεμένοι στην Μαδρίτη ακούσαμε τι είπε η Φόντερ Λάιεν για το Green Deal Πάρα πολύ ωραία αυτή η πράσινη συμφωνία. Υπέροχα Κίνα, η Ιαπωνία, ίσως και οι ΙΠΑ να κάνουν το ίδιο. Όμως τι γίνεται από πλευράς συνομικής μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Ιδάλλως δεν θα γίνει τίποτα. Επίσης, μίλησα και με τον φίλο επίτροπο Νικολά Σμιτ, θα έχουμε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας με το Green Deal αν έχουμε μέχρι το 30 το μισό διοξίδιο, τότε να, σε Φλωρεντία, Παρίσι, στο χωριό μου, στα Πυρηναία, θα πρέπει τα μισά σπίτια να τα μονώσουμε σχολεία, πανεπιστήμια, τις μεταφορές, τη γεωργία, όλα να τα αλλάξουμε. Και τώρα με το βιολογικό αέριο, να χρησιμοποιούμε καλύτερα υλικά και στη γεωργία αυτό βοηθάει την απασχόληση επίσης. Αλλά χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Δεν μπορεί ο κάθε γεωργός να πληρώσει την ε, μόνωση και το κάθε χωριό να μονώσει με δικούς του πόρους στο σχολείο και όταν λέει και παραπέμπει στον Κέννιντι ε, η Φόντερ Λάιεν για το ότι θα κατακτήσουμε το φεγγάρι. Ναι, αλλά μπορεί να μην άρεσε στους λογιστές, αλλά 15 πλάσια άστηκε. Ο προβλήμος της NASA 1,7 δεν γίνεται τίποτα. 400.000 θέσεις απασχόλησης. Με αυτή τη 15 πλασιασμό του προπολισμού της NASA. Και ο Ρούσβελτ έκανε New Deal, αλλά νομίζανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μόνο οικονομική κρίση. Έκανε 15 μεταρρυθμίσεις σε τρει μήνες, πολύ αποτελεσματικό. Και τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός ο ομοσπονδιακός. Ανάλογη φορολογία, χιλιάδες της απασχόλησης, αξιοπρεπής απασχόληση για εκατομμύρια Αμερικανών. Αλλά όμως δεν είναι μόνο λόγια το New Deal. Είναι θέμα προϋπολογισμού και εμείς αυτό θέλουμε στην Επιτροπή μας, παραπέμποντας Ρούσβελτ και Κέννεντ. Τώρα, Green Washing. Επαφή με Τίμερμανς και Φόντερ Λάιν και το επιτελείο τους. Προς το παρόν δεν υπάρχει φρέσκο χρήμα. Να τα ακούει και ο Σαλ Μισελ. 7,7 δις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάθεσης, Μετάβασης. Δεν είναι αρκετά αυτά. Χρειάζεται φρέσκο χρήμα. Αυτό είναι το ένα ρίσκο, δεύτερο ρίσκο. Η νέα χρηματοοικονομική κρίση. Σας ε, απασχολεί αυτό σε επιτροπή, το προβλέπουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι. Σε ένα-δύο χρόνια λένε ότι θα έρθει αλλά εμείς ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή Απασχόληση να το λάβουμε υπόψη. Βλέπετε εδώ το χρέος τον είπα. Είχαμε αύξηση κατά 2,5-3. Βλέπουμε τώρα το χρέος της Κίνας, επίσης ε, ρεκόρ. Ε, το Bloomberg τώρα λέει ότι η επόμενη κρίση θα ξεσπάσει φέτος ή του χρόνου. Έχουμε και τον Τραμπ, αλλά δεν γίνονται πολλά πράγματα. Σαν εσέστερο πλάνο, περίεργο ήχο από τους κινητήρες. Αυτό συμβαίνει τώρα με τη ΣΥΠΑ. Και είδατε τι έγινε με την ανεργία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα περιοριστεί σε ΙΠΑ και Κίνα. Εκατομμύρια ανέργων θα έχουμε. Οπότε πρόκειται για μια προτεραιότητα στη Φοντερ Λάιεν να έχει κάποιο είδου εξασφάλιση, ασφάλεια για την απασχόληση. Τα είπαμε και με τον Νικολά Σμιτ που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για κοινωνικά και μας είπε ότι είναι προτεραιότητα αυτό τη Επιτροπής. Ξέρουμε όλοι ότι έρχεται η κρίση. Θα γίνει στην, την ώρα της θητείας μας θα έχουμε ένα εκατομμύριο ανέργους ή θα κάνουμε κάποιο σύστημα προστασίας. Τα είπε ότι στην Γερμανία υπήρχε ένα πρόγραμμα, ίσως θα πρέπει να κοινοτομήσει και η Ευρώπη ακριβώς όπως έγινε και στη Γερμανία. Αλλά τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Έχουμε πολιετές πλαίσιο και λέμε θα έχουμε σύστημα ασφάλισης εργαζομένων Άρα θα πρέπει να υπάρχει αντίρρησμα στον προπολογισμό. Αυτό αφορά και τη δική σας επιτροπή. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται με το χρέος. Πάρα πολύ ασχήμα τα πράγματα. Όλο ένα και αυξάνει, αλλά βλέπετε ότι σε 30 χρόνια δεν υπήρχε ε, ανάγκη χρέους. Γιατί? Διότι είχαμε κάποιους κοινωνικούς κανόνες και αξίες. Αυτά θέλουμε πριν τον Ρούσβελτ και τους άλλους, πριν τον Μπρέτον Γουτς το καλοκαίρι του 1944. Ο Ρούσβελτ τι έκανε, έφτιαξε τη διακήρυξη της Φιλαδέλφειας, ότι δεν, θέλουμε να, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη κοινωνική χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα, σε όλες τις χώρες και στο παγκοσμίο εμπόριο να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ελάχιστη αμοιβή κλπ. Υπέροχο αυτό το κείμενο. Χωρίς αυτούς τους κανόνες θα έχουμε κρίση, θα έχουμε χρέος. Και μετά, το 1980 τι είπε ο, ο, ο Ρέγκαν, έγινε αυτή η απορρίθμιση, έπεσαν οι μισθοί παντού. Και αυξήθηκε το χρέος το ιδιωτικό και το κρατικό. Ανεξαρτήτως κόμματος όλοι θέλουμε εδώ κοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε επί 30 χρόνια είχαμε ανταγωνισμό, είχαμε ευημερία. Δεν είχαμε χρηματοοικονομική κρίση ούτε χρειαζόταν χρέος γιατί ίσχυαν οι κοινωνικοί κανόνες. Μόλι τους απεμπολίσαμε τότε είχαμε πιο ευάλωτη απασχόληση και όλοι επλήξαν στην καθημερινή τους ζωή. Για όλους αυτούς τους λόγους σας λέω ότι ο προπολογισμό του 2021 είναι το θέμα του πολιτού πλαισίου και το τι θα γίνει και με, το, με τη νέα συμφωνία, το New Green Deal, εν αποτελεσματικότητα της ενέργειας. Και γι' αυτό και ευτυχώς που τα λέμε σήμερα, γιατί θα πρέπει να, ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα. Πώς θα έχουμε ένα σύστημα προχωρημένο για την εξασφάλιση των εργαζομένων και πάλι συμπαθάτε με που δεν έρχομαι συχνά εδώ, αλλά είναι θέμα χρονοδιαγράμματος. Ο Σαλουτσέλη θα το κλείσει το Φεβρουάριο, δεν τον πιστεύει κανείς. Αλλά τουλάχιστον να πάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και εμείς στην Επιτροπή των Προπολογισμών επίσης να κάνουμε ό,τι χρειάζεται οι ίδιοι ακροάσεις, να απεμπλοκεί η διαδικασία. Ξέρουμε ότι δεν θα δώσει ούτε η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ελλάδα, ε, συγγνώμη, η ε, Γαλλία, η Γερμανία το ένα δις που χρειάζεται. Άρα κοινωνική δικαιοσύνη για όλους και φορολογική δικαιοσύνη και για τους νέους. Όμως εμείς δεν θα μπούμε στα χωράφια σας. Εσείς η δική σας επιτροπή να προστατεύσει την απασχόληση. Γι' αυτό θέλουμε η κάθε επιτροπή να ασχοληθεί με τα δικά της, τι θα γίνει δηλαδή με μεταφορές κλπ. κλπ. Αυτά, Πρόεδρε, έχω άλλο χρόνο ή όχι. Έχουμε, λέει ο Πρόεδρος. Τρία, τρία έχετε, τρία λεπτά έχετε. Α, καταλαβαίνετε και τα γαλλικά. Σας ευχαριστώ. Το λέει και η Κομισιόν. Φτιάξει 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση. Πολύ σημαντικό. Όλοι οι δήμαρχοι. Έχουμε 10.000 μικρά χωριά που έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα και λένε για απασχόληση και στα μικρά χωριά. Είχα πάει στην Κρενόβλα, έλεγε κάποιος για την μόνωση, δεν έχω πολλά λεφτά, μεσοεργατική κατοικία. Και έχω 800 ευρώ το χρόνο παραπάνω με την ε, μόνωση. Παντού θα ισχύσει το ίδιο. Αλλά μπορώ να ε, βοηθήσω, έλεγε ο Δήμαρχος της μόνο τρία σπίτια το χρόνο. Δεν έχω χρήματα από την Ευρώπη, Άρα αυτό χρειάζεται. Να έχουμε θέσει απασχόληση, να μην έχουμε εγκαταστάσει, αγοραστική δύναμη. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Έχουμε αυτό το έγγραφο της 14ης ε, Ιανουαρίου της Επιτροπής και λέει εδώ ότι χρειάζονται 600 δις ετησίως και για, για αυτή την μόνωση. Άρα θα πρέπει αυτά να τα διαπραγματευτούμε. Επίσης ε, χρειάζεται να μας δώσουν άλλα 16 δις για να έχουμε τη σωστή μόχλευση σε κάθε κλάδο. Θα πρέπει να δούμε τι λειτουργεί καλά και τι όχι, που δημιουργείται απασχόληση, που υπάρχει αποτελεσματικότητα, να έχουμε νέα μέσα πολιτικής δεν υπάρχει μαγικό ρευδάκι, χρειάζεται χρηματοδότηση. Άρα εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερο προπολογισμό με ιδίους πόρους, να μην θυγούν οι φτωχότεροι, 30% Πολωνών, Γάλλων, ε, μπαίνουν μέσα, είναι στο κόκκινο, κάθε μήνα. Και για το κλίμα, να δούμε τι μπορεί να γίνει, όσον αφορά την τράπεζα για το κλίμα. 16 δις κάθε χρόνο θα είναι τα, τα δάνεια. Αλλιώς δεν αρκούν τα χρήματα που δίνονται. Αλλά και η κεντρική τράπεζα θα δώσει 240 δις φέτος. Οπότε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Οικονομική Επιτροπή θα δούμε πως θα έχουμε καλύτερο προϋπολογισμό γιατί έχουμε 600 δις διαθέσιμα κάθε μήνα στην Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα χρήματα, αντί να βγαίνουν σε κερδοσκοπία, να πάνε για απασχόληση και για την κλιματική τράπεζα. Επομένως, να έχουμε νέους πόρους, να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νέες λύσεις καλύτερος προϋπολογισμός είναι οι διάφοροι φόροι για άνθρακα στα σύνορα, για πλαστικό κλπ. Φορολογική δικαιοσύνη, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της ενδοευρωπαϊκής ε, κρίσης φορολογικού ανταγωνισμού. 45% βλέπουμε εδώ, χρειάζονται 19% φόρου κερδών. Τώρα έχουμε τα μερίσματα και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Πού πάνε τα κέρδη, πάνε στους εργαζομένους ή πάνε σε επενδύσεις για το μέλλον ή φεύγουν από την πραγματική οικονομία. Όσα δεν επανεπενδύονται από κανέναν και πάνε στις αγορές, αυτό είναι πρόβλημα μακροοικονομικό όλο ένα περισσότερα μερίσματα και όλο ένα και λιγότερο φόρο στα κέρδη. Αυτό δεν είναι New Deal, δεν είναι τι είπε ο Ρούσβελτ. Είχαν ρίξει τους φόρους πάρα πολλές ε, ε πολιτείες τότε, αλλά μέσα σε τέσσερις ε, μήνες είπε όλοι θα έχουν 38% σε όλες τις πολιτείες. Είδατε τι γίνεται στις ε, είπα, ε, ε, Ήταν 38% επίρους βελτοφόρος και, και δεν μιλάμε για την Σοβιετική Ένωση, το αντίθετο. Άρα υπήρχε ομοσπονδιακός φόρος 38% επί των κερδών και εμείς έχουμε 19% σχεδόν τα, τα μισά. Οπότε, το προπολογισμό λέει να έχουμε έναν φόρο επί των κερδών δεν θα θίξει τους βιοτέχνες της μικρές επιχειρήσεις. Αλλά αν θέλουμε ιδίου πόρους, φιλόδοξο προϋπολογισμό, θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Καλύτερος προϋπολογισμός θα μπορούσε να βοηθήσει το κόστος διαδίω για κάθε χωριό, για κάθε οικογένεια, για κάθε επιχείρηση να υπάρχει ενίσχυση και το μισό να χρηματοδοτείται από την και ε, με αυτή την έννοια θα είναι χρήσιμη η Ευρώπη. Δεν έχω βέβαια χρόνο ε, να αναπτύξω. Φαίνεται ότι από ό,τι καταλαβαίνω έχω ξεπεράσει και το χρόνο ε, εργασίας. Θα σας στείλω, ομιλία, συγγνώμη, θα σας στείλω όλα τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την εξαιρετική σας παρουσίαση. Και τώρα θα τα πω τσέχικα όμως. Και θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Ναι, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε χρόνο, δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τα πάντα. Ωστόσο, νομίζω ότι αν είμαστε όλοι τυπικοί, ίσως θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για αρκετά θέματα και να δούμε τον προϋπολογισμό από την πλευρά του, ε, της ε, ΕΜΠΛ. θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια ε, πληρωμές για το 2021 ε, αυτές θα εστιαστούν στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων ε, από το, 20, από το 14 στο 20 νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει ε, πρόσκομα για δημιουργία νέων προγραμμάτων και δεν θα πρέπει να γίνει ε, τη ζημία το, του κοινωνικού ταμείου όπως έγινε στο παρελθόν εκτός από το ESF Plus πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και την υποστήριξη άλλων εργαλείων όπως ας πούμε European Globalization Fund Fund, ε, βοήθεια για τους Ταμείο για τη Βοήθεια των Φτωχοτέρων κλπ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βέβαια για όσα μας είπατε. Ε, θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω και την σημασία των πολιτικών προγραμμάτων ε, στην προετοιμασία του προϋπολογισμού. Ίσως τα ποσά να ακούγονται ε, μικρά, αλλά μπορούν να αποτελέσουν όταν προετοιμάζονται με προσοχή, να αποτελέσουν, λέω, καινοτόμε λύσεις για πολλά θέματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα από το παρελθόν ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, που υλοποιήθηκε από την Κομισιόν και που μετά έγινε ε, κεντρικό στοιχείο της πολιτικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Θέλουμε τα πιλωτικά προγράμματα να αξιολογούνται και να βασίζονται σε πραγματική προστιθέμενη αξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Επιτροπή και τις Γενικές Διευθύνσεις καθώς επίσης και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, πέρσι μαζί με τον Πέτρο Πόλα και είχαμε υποβάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα σχετικά με την ε, κοινωνική στέγαση των ε, Ρωμά. Ήταν, ενδιαφέρθηκε η Κομισιόν στην υλοποίηση του προγράμματος, αλλά μειώθηκε κατά 50% περιακόπη δηλαδή από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και έτσι η υλοποίηση κατέστη αδύνατη. Τα, το πολιτικό πρόγραμμα λοιπόν περιορίστηκε σε μία χώρα αντί για τις αρχικές τρεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε εμείς θα ζητήσουμε να ε, ε, επανυποβληθεί το πρόγραμμα αυτό και θέλουμε να το προωθήσουμε το πρόγραμμα αυτό φέτος. Επίσης ε, θα συζητήσουμε αργότερα και άλλα θέματα. Αυτό ήταν απλώς ένα ξεκίνημα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους άλλους σκιώδεις σοσιαλιστές Μάρκα Ίντζελ, πώς το λέτε το όνομά σας, δεν βαριέστε όπως να είναι. Θα ήθελα να μιλήσω στο όνομα του κύριου Ελισεκ Μίλλερ, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τους προβληματισμούς της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο της έκθεσης, ευθυγραμμίζεται με ε, τις προτεραιότητές μας. Αναφέρεται για παράδειγμα στο φρέσκο χρήμα ε, για τις δράσεις αυτές ε, και όχι να γίνει εις βάρος ε, άλλων γραμμών του προπολογισμού αναφέρεται στη δίκαιη μετάβαση. Επίσης, ε, επιμένουμε στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Χρειάζονται λοιπόν επαρκή πόροι, ιδιαίτερα για την δημιουργία της εγγύσης για τα παιδιά. Επίσης, σημαντικό είναι στο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, στις διαπραγματεύσεις αυτές, ε, να συμπεριλαφθεί και το ESF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ είναι σημαντικό να έχουμε φιλόδοξο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς καθυστέρηση, με ισχυρό επίκεντρο στην κοινωνική πολιτική, να έχουμε ένα ισχυρό ταμείο δίκαιης μετάβασης με αρκετή χρηματοδότηση, ώστε να μην παίρνει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι ήδη αρκετά δύσκολη η κατάσταση και επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας διότι οι τροπολογίες ε, και οι συνεισφορές της ε, Επιτροπής μας ε, δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Ευχαριστώ πολύ για τις συγκεκριμένες προτάσεις σας. Δίνω το λόγο στην Σαμίρα Ραφαέλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και την εισηγήτρια. Ήταν πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα αλλά είναι πολύ θετικό το ότι μπορούμε να ε, δώσουμε και τη δική μας συνεισφορά στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα που άπτεται και των δικών μας εργασιών. Ε, είχαμε αρκετές προτάσεις και από το ΡΙΝΙΟΥ. Νομίζω ότι το βασικό κλειδί είναι να τονίσουμε την ε, σημασία μιας κοινωνικής Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Σημαντικό εδώ λοιπόν είναι να προωθήσουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και να εντοπίσουμε τα κενά στον προϋπολογισμό, τα σημεία όπου μπορεί να υπάρξει αποκλεισμό στον προϋπολογισμό αυτών. Υπό αυτή την προοπτική λοιπόν εξετάσαμε το θέμα και κάποιες από τις τροπολογίες που ήθελα να τονίσω είναι για παράδειγμα οι τροπολογίες για τις πολιτικές που προωθούν μια ε, κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και μέτρα που προωθούν την ισότητα και την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας για άντρες και γυναίκες. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρουν ε, προτάσεις που λένε ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που κινδυνεύει από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να έχει πρόσβαση στα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και Κάτι που συχνά παραβλέπεται είναι η ε, πόροι για ε, τα υπερπόντια ε, εδάφη. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα τα υπερπόντια εδάφη που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα όσον αφορά τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πραγματικούς ε, πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στη σωστή μετάβαση. Από πλευράς του Ρινιού, λοιπόν, εξετάσαμε πού μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερη αξία για να έχουμε ε, μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν από το ID. Ούτε βλέπω την κυρία Μαρία Πετερχάνσεν. Θα δώσω το λόγο στην Σάντρα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αυτή τη στιγμή που δεν έχει καθοριστεί ακόμα το πολιτεύσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να προωθήσουμε την ε, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Αυτό είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν, δεν επιτρέπεται να αποκλείσουμε τους φτωχούς Ευρωπαίους πολίτες από την εξίσωση. Εξετάσαμε τα εργασιακά δικαιώματα, την στέγαση σε προηγούμενες εκθέσεις μας. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι θέματα υψίστης σημασίας. Αυτό που έλειπε από την μελέτη της Eurofund ε, για τις επισφαλείς θέσεις εργασίας και ε, την φτώχεια είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει επαρκές εισόδημα. Κυρίως ε, κινδυνεύουν ε, από τη φτώχεια οι γυναίκες, ε, οι άνθρωποι με μερική απασχόληση, οι γεωργοί, οι άνθρωποι με επισφαλείς οικογενειακές σχέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι ακόμη πιο ευάλωτοι στις καταστάσεις που περιγράψατε εσείς. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε μία έκθεση χωρίς ενίσχυση της εδαφικής και της κοινωνικής συνοχής τη στιγμή που έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός για ε, δαπάνες στην άμυνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε το λόγο? Όχι, ωραία. Εάν όχι, θα ρωτήσω τον εισηγητή εάν θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην πρώτη σας ανησυχία. Αν βρισκόμαστε σε κρίση ε, πληρωμών, ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε το 2021 έχουμε 184 ε, πιστός πληρωμών, πράγμα που θα μας επιτρέψει την αποφυγή της κρίσης που είχαμε πριν από 7 χρόνια. Έχουμε ένα συν 2, ένα συν 3. Γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε στη νομική βάση και θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε ε, προσεκτικά. Ε, ε, προσέχουμε λοιπόν και υπάρχει το έγγραφο των guidelines το οποίο είναι πάρα πολύ σύντομο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα, αλλά πάντως ε, επιμείναμε πάνω σε αυτό, καθώς επίσης και για τα PPA, τα οποία είναι πολύ συχνά καινοτόμα προγράμματα. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούν προβλήματα. Κοιτάξτε, ούτω ή άλλω εγώ, όπω σα είπα και στην αρχή, εδώ και έξι μήνε είμαι βουλευτή, δεν φέρνω όλε τι αμαρτίε του παρελθόντο. Απ' την άλλη πλευρά όμω, είναι γεγονό ότι είναι δύσκολο. Ε, υπάρχουν βουλευτέ, πολλοί βουλευτέ, οι οποίοι ε, ε υποβάλλουν ε, πολλέ PPA που είναι δηλαδή αυτέ τι συνεργασίε ιδιωτικού και δημόσιου ε, και είναι δύσκολο να κάνουμε το ξεκαθάρισμα ε, για να μας ε, βοηθήσετε και για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε στο ξεδιάλεγμα θα πρέπει να μας δίνετε πραγματικά πολλά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών και γι' αυτό ακριβώς βρίσκομαι σήμερα εδώ θέλει να συνεργαστεί μαζί σας ε, και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι πρέπει όλοι στο Κοινοβούλιο να δουλέψουμε. Σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Μάρκ Άντζελ, το θέμα του κοινωνικού πυλώνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ε, δεν ενδιαφερόμαστε για έναν προπολογισμό ο οποίο θα κόβει από τον ένα για να δίνει στον άλλον και θα κόβει από τον άλλον για να δίνει στον τρίτο. Ε, αυτό που θέλουμε δεν είναι να μην αγγίξουμε τίποτα, αλλά θέλουμε μια πραγματική Ευρώπη και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να ε, δουλεύει ας πούμε υπέρ του κλίματος ε, περικόπτοντας τον προϋπολογισμό για τη γεωργία και τελικά να αυτοκτονούν ας πούμε οι γεωργοί γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Ε, το γεγονός ότι σταματούν ας πούμε οι ποσοστώσεις γάλακτος δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε τους γεωργούς στη Γαλλία, στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού ε, και ε, ε, είναι γεγονός ότι με τις ποσοστώσεις ειδικά από ζούσαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι από την δουλειά τους ακόμα και σε ορεινές περιοχές δεν χρειαζόντουσαν επιδοτήσεις γιατί μπορούσαν να ζήσουν από την δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αν καταραίει το σύστημα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουν δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ε, θέλουμε να μείνουν οι γεωργοί στις ε, δουλειές τους, θα πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε. Ε, επίσης υπάρχουν ειδικέ καταστάσεις στη Γαλλία, στο Βέλγιο, μείον 30% ε, λόγω των ε, πλημμυρών χάθηκαν από τα σιτηρά. Επίσης στην Πολωνία ας πούμε υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα όσον αφορά άλλες παραγωγές. Όταν από τη μία μεριά λέμε στον Γεωργό πρέπει τώρα να παράγεις βιοαέριο θα πρέπει να τον βοηθήσουμε σε αυτό το μετασχηματισμό. Ε, στην Ευρώπη πολύ σημαντικό είναι να έχουμε μια ιδέα ε, σωστή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και από την άλλη μεριά, ε, βεβαίω, ναι, όλοι μα κοιτούν, στρέφονται προ εμά για να δουν τι θα κάνουμε όσον αφορά το κλίμα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην σταθούμε στο ύψο μα και όσον αφορά τα κοινωνικά. Και πραγματικά δεν τίθεται κανένα ζήτημα λόγω του περιβάλλοντο να υπονομεύσουμε την κοινωνική διάσταση. Ε, απ' την άλλη πλευρά, συγγνώμη αν ε, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν ε, προώθησε κάποια από τα προγράμματά σας. Από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι 60% των βουλευτών μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι νέοι βουλευτές ε, και επομένως νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε νέους πόρους. Το Κοινοβούλιο είχε πει ότι δεν θα μπορέσει να ψηφίσει το νέο ΠΔΠ εάν δεν έχει προχωρήσει το θέμα των ιδίων πόρων. Ε, και αυτό ε, ήταν πριν από την Πράσινη Συμφωνία. Αν θέλουμε τώρα χρηματοδότηση και για τον Green Deal και για την Πράσινη Συμφωνία, θα πρέπει οπωσδήποτε πραγματικά να έχουμε ε, νέους πόρους. Θα πρέπει να αυξηθούν οι ίδιοι οι πόροι και ενδεχομένως να βρούμε και πόρους μη δημοσιονομικούς το, στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, ο Μπαράκ Ομπάμα πέρασε το νόμο του όσον αφορά ε, ε, έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα. Ίσως θα πρέπει να βρούμε έναν νόμο φάτκα κλίματος. Εγώ δεν μιλάω τώρα σαν εκπρόσωπο του προπολογισμών, αλλά θα πρέπει να δούμε πραγματικά τι θα γίνει με του ίδιου πόρου και να δούμε, ε, να δούμε τι θα γίνει. Ε, έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ακούει και είναι μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει η συζήτηση αυτή. Ε, σχετικά με αυτό που έλεγε η κυρία Ραφαέλα για την ε, ε, Ευρώπη η οποία περιλαμβάνει όλο τον κόσμο, δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο. Το θέμα επίσης που έθιξε η Σάντρα Περέιρα δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να λέμε «Α, τι κρίμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, ψήφισαν κατά της Ευρώπης, ας πούμε, σε εκλογές», αλλά από την άλλη μεριά ε, και η Ευρώπη θα πρέπει να ε, δείξει, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τον προϋπολογισμό και με τις πράξεις, ότι πραγματικά υποστηρίζει τους πολίτες. Δεν μπορεί να λέμε «Α, δεν αγαπάνε οι πολίτες στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη να μην κάνει τίποτα για τις για, τη, για τους ε, πολίτες. Ε, το Λουξεμβούργο έχει δείξει μια, αυτό το μακροχρόνιο ε, δρόμο που οδηγεί σε μεγαλύτερη ευημερία με μηδέν ανεργία. Άρα πρέπει προς τα εκεί να προχωρήσουμε. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια συμπεριληπτική Ευρώπη η οποία να λαμβάνει όλους τους πολίτες υπόψη όσον αφορά την αγοραστική δύναμη και θα τελειώσω με αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να σταματήσουμε με αυτές τις μικρές δουλίτσες ε, με 400-450 ευρώ. Ε, είναι πραγματικά καταστροφικές τέτοιου είδους ε, δουλειές. Επομένως, ναι, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την αστάθεια. Επίσης, όταν λέμε, ας πούμε πρέπει να σας πω ότι ε, ένας άνθρωπος ε, ο οποίος ζει σε, ένα καλό σπίτι, που ζει σε ένα καλά ε, μονομένο σπίτι και ο οποίος λέει ότι 800 ευρώ έχω κερδίσει από τον λογαριασμό της ενέργειας και δεν το λέει ένας ευρωβουλευτής ή κάποιος που δουλεύει στην Κομισιόν, ένας απλός άνθρωπος που λέει κέρδισε 800 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα θα πρέπει να πείσουμε και την Κεντρική Τράπεζα να δώσει χρήματα γι' αυτό. Ε, ζητώ συγγνώμη που μακρύγω αλλά και το θέμα των ε, κατευθυντηρίων γραμμών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον Ιούνιο η Κομισιόν ε, θα μας ε, υποβάλει ένα πρώτο σχέδιο και επομένως τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην ΕΜΠΛ θα πραγματοποιηθεί 20 Φεβρουαρίου. Τροπολογία στην ε, ε, ψηφοφορία στις 30 Μαρτίου στην Επιτυσσουσίας Αρμόδια Επιτροπή και στην Ολομέλεια θα πάει τον Απρίλιο του 2020. Συνάδελφοι, αυτό ήταν το τελευταίο θέμα στην ημέρηση διάταξή μας. Θα ήθελα απλά να σας πω ότι 18 Φεβρουαρίου θα είναι η επόμενη συνεδρίαση από τις... 5 και 4 έω τι 7, 20 Φεβρουαρίου από τι 9 στις 12.30 στις Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου από τις 3 έω τι 6.30 στις Βρυξέλλες και 17 Μαρτίου του 2020 από τι 9 έως τις 12.30 και από τις 2.30 έως τις 6.30 και πάλι στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ θερμά. Και δεν ξέρω αν σας είπε κανείς ότι σας αγαπάει κανείς την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εγώ όμως σας αγαπάω. Ε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας στην Προεδρία μου. Πρώτη φορά προείδρευσα. Ελπίζω να μην τα πήγα και πάρα πολύ άσχημα. Σας εύχομαι ότι καλύτερο. Καλό βράδυ και ο Πρόεδρος ευχαριστεί θερμά και τους διερμηνείς και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστεί και το προσωπικό της Επιτροπής Απασχόλησης, τους συναδέρφους, τους εισηγητές, όλους. Καλό βράδυ σας εύχομαι και να χαμογελάτε. Καλό σας βράδυ.